Ladies and gentlemen, good afternoon. Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ. Θα αρχίσουμε αμέσως, αν και καθυστερήσαμε λίγο, τώρα έχει έρθει ο συγγετής μας για να συζητήσουμε την έκθεση για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση που ανέλαβε η ΣΕΝΤΕ από κοινή πρωτοβουλία της ΑΦΚΟ και της ΑΦΕΤ Η μετά τη σύσκεψη των συντονιστών, ε, οι φιλελεύθεροι ανέλαβαν την έκθεση. Και θα ακούσουμε την, ε, την πρώτη παρουσίαση του σχεδίου έκθεσης από τον κύριο Ούρμα Σπάιτ. Ναι, λίγο ασυνήθιστο το χρονοδιάγραμμα γιατί συνεδρίασή μας. Θα ακολουθήσουμε την συνήθεια διαδικασία. Πρωτού περάσουμε στην έκθεση. Θέλω να θυμίσω ότι αναμεταδίδεται η συνεδρίασή μας στο διαδίκτυο. Φυσικά τα τακτικά μέλη έχουν προτεραιότητα για τη διερμηνία. Θα ήθελα να εγκρίνουμε το σχέδιο μέσης διάταξης απουσία ενστάσεων ε, θεωρώ γεκριμένη τη μέσα διάταξη. Ανακοινώσει της Προέδρου τώρα. Έχει πάρα πολύ περιορισμένο χρόνο ο κ. για την παρουσίασή του και γι' αυτό θα ήθελα το ταχύτερο δυνατόν να αρχίσουμε. Έχει αποφασιστεί από την Επιτροπή Ελέγχου των Προϋπολογισμών από την Επιτροπή ΙΜΚΟ και ΑΦΚΟ. Τρεις νομοδοτήσεις έχουν αποφασιστεί λοιπόν για αυτή την έκθεση. Ο κ. Γκονζάλες Πόνς είναι ο εισηγητής νομοδότησης της Επιτροπής προϋπολογισμών. Τέβιτ Μακάλιστε για την Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων και Λάρα Κόμη για την ΕΜΚΟ. Χωρίς ε, περαιτέρω καθυστέρηση, δίνω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Πάτ. Παρακαλώ, παρουσιάστε μας το σχέδιό σας. Ευχαριστώ, Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, το άρθρο 42 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση απαιτεί τον προοδευτικό προσδιορισμό της Κοινή αμυντικής πολιτικής ένωσης στο πλαίσιο της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας, η οποία θα οδηγήσει σε μια κοινή άμυνα όταν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο λάβει σχετική απόφαση. Το ίδιο άρθρο προβλέπει τη δημιουργία των δύο θεσμών άμυνας, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και της, της ΠΕΣΚΟ, του Μόνιμης Διαρθρωτικής Συνεργασίας, καθώς και τον προσδιορισμό ε, της ε, μάχημης ικανότητας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, θα πρέπει να υπάρχει συμβατότητα με τον ΝΑΤΟ και αμοιβαία υποστήριξη όλα τα στοιχεία προς την συγκρότηση του Εθνικού Οργανισμού του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Αμήνης έχουν υλοποιηθεί. Ο σταδιακός προσδιορισμός της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης θα μας οδηγήσει στην ένταξή του στο επόμενο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και επίσης θα εκπονηθεί η διαδικασία σε σχέση με το τι έπεται για τα θέματα Ασφάλεια και άμυνα ε, για το εκτελεστικό σχέδιο για αμυντικά ζητήματα ε, και μια πιθανή Ευρωπαϊκή Λευκή Βίβλο για το ζήτημα για την, ε, και για την περιγραφή των παρασκευαστικών δράσεων που θα πρέπει άμεσα να δρομολογηθούν. το αμυντικό περιβάλλον έχει αλλάξει με ραγδαίους ρυθμούς τα τελευταία χρόνια και θα πρέπει να αλλάξουμε το ευρωπαϊκό μοντέλο ε, ενεργοποιώντας πλήρως το άρθρο 42 της ε, συνθήκης. Ε, μέχρι στιγμής η διάσταση άμυνας Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι κενέ δηλώσεις επί της αρχής προς το παρόν. Ακόμη δεν έχει αναπτυχθεί ευρωπαϊκός οργανισμός και οι μάχημες ομάδες ακόμη δεν έχουν χρησιμοποιηθεί στην πράξη. Μετά τις επιθέσεις στο Παρίσι η, η Γαλλία ήταν η πρώτη που Επικαλέστηκε το άρθρο 42,7 για την αρρωγή. Οι επιπτώσεις ε, των τρομοκρατικών επιθέσεων στο Παρίσι και μετά των επιθέσεων, της επίθεσης στις Βρυξέλλες οδηγούν σε μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση ότι διακυβεύεται η ασφάλεια στην Ένωση. Σήμερα η πλειοψηφία των πολιτών μας υποστηρίζουν μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση τον επομιστό την ευθύνη σύνταξη τη έκθεση ε, του Κοινοβουλίου για την Ένωση ε, αποφασίζω να ζητώ, ζητήσω από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να αρχίσει τον προσδιορισμό τη Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση σε βάση το 42 τη Συνθήκη. Επίση, θέλουμε να συγκροτηθεί μόνιμη ομάδα εργασία υπό την αιγίδα τη ΕΙΠΑ τη εκπροσώπου και με συμμετοχή των κρατών μελών προτείνουμε δε σταδιακή προσέγγιση. Ε, διαβλέπουμε ανάγκη εντατικότερη συνεργασία ανάμεσα στα κράτη-μέλη ε, και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνα μέσα από τη Διευθυντική Συνεργασία ΠΕΣΚΟ και με τη συγκρότηση διεθνών ομάδων στα πλαίσια τη ΠΕΣΚΟ ε, και θα τεθούν στην υπηρεσία τη κοινή πολιτική ασφάλεια και άμυνα. Παραδείγματο χάρη σε αυτή τη λογική τη ευφυού προσέγγιση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, το πρώτο βήμα θα είναι η πρώτη ε, πολιτική για την μάχη μη δυνατότητα και για τον εξοπλισμό, καθώ και την έρευνα για τον αμυντικό εξοπλισμό, τόσο να μεγιστοποιήσουμε τα ωφέλη των κονδυλίων διαθέτουμε. Επιθυμούμε προδραστική συνεργασία ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ ε, ενισχύοντα την ανθεκτικότητά μα, ε, κυρίω στο Νότο και στην Ανατολή, υποστηρίζοντα τα διεθνή τάγματα στα κράτη-μέλη, κυρίω στο Ανατολικό μέτωπο, ε, η συνεργασία με τον ΝΑΤΟ θα πρέπει να ενισχυθεί. Δεν σημαίνει αυτό ότι ο ρόλο του ΝΑΤΟ ε, υποβιβάζεται. Θα πρέπει να εμβαθυνθεί η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά είναι συμπληρωματικό ο ρόλο. Επιθυμούμε τη συνέργεια και με πλήρη σεβασμό του θεσμικού πλαισίου ε, κατά την, ε, και διατηρώντα την αυτονομία ω προ τη λήψη αποφάσεων για τα δύο μέρη. Η σχέση των δύο θεσμών θα πρέπει να οδηγήσει ε, σε ενίσχυση ανταγωνιστικότητα τη Ευρωπαϊκή Ένωση και στην ενίσχυση των διατλαντικών σχέσεων με τη ΣΥΠΑ και με τον Καναδά. Επίσης, θα πρέπει να έχουμε ένα ευρωπαϊκό σύστημα για την ε, ταχεία εξέλιξη των, ε, του προσωπικού και του εξοπλισμού. Είναι ένας χώρος ε, όπου προτείνουμε δραστική μείωση τη γραφειοκρατία, ε, ούτω ώστε οι μάχη ομάδε να μετακινούνται ε, χωρί καθυστέρηση όταν συντρέχει ανάγκη. Και θα ήθελα να αναφερθώ επίση στην ανάγκη να αναπτύξουμε μια διαδικασία επί ε, τη βάση τη διετή χρήση, ούτω ώστε να αναπτυχθεί και ευρωπαϊκή νομοθεσία σε αυτό το τομέα. Επίση, για την Μελλοντική Αμυντική Ένωση ως προς τον προϋπολογισμό ζητούμε το 2% στόχο του ΕΠ και από τα πλευρά των, των κρατών μελών και το 20% ε, για αυτά για την έρευνα. Επίσης πιστεύουμε ότι μπορούμε να έχουμε ε, υποδομές όπως ε, γέφυρες ε, και οδικά δίκτυα που θα βοηθήσουν τα κράτη-μέλη σε αυτή τη δράση στο μέλλον. Το Σεπτέμβριο του 2013 οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων ζήτησαν προπαρασκευαστική δράση για την έρευνα στον τομέα της αμυντικής βιομηχανίας ε, και αυτό το ζητήθηκε εξάλλου από την θέση σε ισχύ τη συνθήκη Λισαβόνα. Χρειαζόμαστε καλύτερε και περισσότερε επενδύσει και καθώ και συνεργασία στον τομέα τη ε, έρευνα ε, τη αμυντική βιομηχανία. Η ύπατη εκπρόσωπο, η κυρία Μοκερίνη, παρουσίασε με τον Ιούνι μια ευρωπαϊκή στρατηγική για την αμυντική διάσταση όπου τονίζει ότι χρειαζόμαστε μια πιο διαστρωμένη συνεργασία, επενδύσεις για την έρευνα και την τεχνολογία και μια ε, κρατεότερη εσωτερική αγορά, εφοδιαστική ασφάλεια και προστασία ε, της ε, βιομηχανικής και τεχνολογικής βάσης για τον αμυντικό εξοπλισμό. Καλό είναι, προβλέπει είπατε ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπος ένα συνολικό σχέδιο ε, και το, στην, Πρατι, στην Πρατισλάβα αναφέρθηκε αυτό στο, στη Σύνοδο στο Σεπτέμβριο, αλλά μην ξεχνάμε ότι μας λείπει η Λευκή Βίβλος που θα επέτρεπε να έχουμε μια συνολική στρατηγική για να δούμε ποια θα είναι ή πώς θα ενταχθεί μάλλον ε, ε, η Αμυντική Ένωση στο επόμενο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο. Ο πρόεδρος Γιούγκερ στην φετινή του ομιλία επικεντρώθηκε στην αμυντική πολιτική ε, και αναφέρθηκε στην ανάγκη μάχημων ομάδων για στρατιωτικές επιχειρήσεις, στην ανάγκη διαρθρωτικής μόνιμη συνεργασίας και πρέπει να επενδύσουμε στην έρευνα και στην καινοτομία Μας προ τον αμυντικό εξοπλισμό. Περιμένουμε το σχέδιο δράση δε μέχρι το τέλο του τρέχοντο. Στη Σύνοδο στην Πρατισλάβη, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων δήλωσαν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να ισχύσει τι προσπάθειέ τη ω προ την αμερική πολιτική, ακολουθώντα τη γραμμή του Προέδρου Γιούγκερ. Η Γερμανία και η Γαλλία επίση έχουν εκφράσει ε, τι ε, σαφέστατα τι απόψει του για την ενίσχυση τη αμυντική ε, πρόσφατα. Οπότε, υπό το φω των εξελίξεων στον τομέα αυτό, νομίζω υπάρχει ο κατάλληλο δυναμικό για να προωθήσουμε την αμυντική πολιτική ενισχύοντας το ε, σε συμπληρωματικό ρόλο ως προς τον ΝΑΤΟ, προστατεύοντας τα ευρωπαϊκά συμφέροντα και τον τρόπο ζωής μας. Για το χρονοδιάγραμμα, για τις τροπολογίες για τις έκθεσεις. Ε, είχαμε την 7η Σεπτεμβρίου, 7 Σεπτεμβρίου ως ε, καταληκτική ημερομηνία. Ήταν πολύ άριθμες τροπολογίες, ε, θα τις εξετάσουμε. Στις 12 ή 10 Οκτωβρίου θα γίνει η δεύτερη εξέταση του σχεδίου έκθεσης και αναμένεται το Νοέμβρη στην Ολομέλεια να περάσει η έκθεση από το σώμα. Τέλος θα πρέπει να δράξουμε την ευκαιρία και να μεταλλευτούμε αυτό το δυναμικό που υπάρχει για να ενισχύσουμε την Αμυντική Ένωση και δεν θα πρέπει να ε, χάσουμε αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Βρίσκω μια διοργάνωση αυτής της συζήτησης. Αναγνωρίζω έναν από τους ε, συντάκτες της ε, έκθεσης τον κύριο Μακάλιστερ, ε, που είναι μέλος της ΑΦΚΟ. Θέλετε να πάρει το λόγο, κύριε Μακάλιστερ. Ναι, αν συμφωνούν και οι άλλοι, να πω και εγώ δύο λόγια. Μου ζήτησε η Επιτροπή ΑΦΚΟ να ετοιμάσω μια γνωμοδότηση. Η συνάντηση για να ολοκληρώσουμε την ε, γνωμοδότηση με τους κοιόδης εισηγητές αρχικά είχε, είχε προγραμματιστεί για σήμερα το απόγευμα, αλλά τελικά ε, θα αναβληθεί και τώρα είμαστε στη φάση της γραπτής διαδικασίας. Στις προτάσεις που έκανα ε, υπάρχουν 7 σημεία όπου κάνω συγκεκριμένες υποδείξεις για το πώς θα εντάξουμε, πώς θα ενσωματώσουμε κάποια σημεία στο ψήφισμα αυτό. Καταρχάς, υπενθυμίζουμε ότι η ΚΠΑ, όπως προβλέπει η συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα πρέπει να ε, έχει μια προοδευτική πλαισίωση μια κοινή αμυντικής ε, πολιτικής. Δεύτερον, ε, για να ειδοποιήσουμε τους στόχους της ΚΠΑ, θα πρέπει να ενισχύσουμε το επιχειρηματικό δυναμικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να δρά προς το εξωτερικό, για αποτροπή των συγκρούσεων, ε, ε αποστολές κτλ. Ε, γιατί το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείται η Ευρωπαϊκή Ένωση ασφάλειας είναι όλο και πιο έντονα επιδεινούμενο. Επίση, ζητάμε από την ΥΠΑΤΕ εκπρόσωπο και τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν το δυναμικό τη Ευρωπαϊκή Συνθήκη, ιδίω το άρθρο 44 για την εφαρμογή τη ΚΠΑ, και το άρθρο 46 για τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία για να υπάρξει μια πιο γρήγορη και ευέλικτη ανάπτυξη των αποστολών ΚΠΑ ε, και των επιχειρήσεων της ΚΠΑ. Τέταρτον, ζητάμε το Συμβούλιο, την Κομισιόν και την ε, Αντιπρόεδρο και είπα πρόσωπο εκπρόσωπο να εξασφαλίσει αυτό που προβλέπει η συνθήκη ε, ότι θα υπάρχει μια συνέργεια μεταξύ των διαφόρων τομέων μέσω μιας συνεκτικής προσέγγισης. Πέμπτον, να δημιουργηθεί ένα μόρφωμα του Συμβουλίου με τους Υπουργούς Άμυνας, με μια επιχειρησιακή διάσταση. Ε, επίσης, ε, θα πρέπει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας να έχει και επιχειρησιακό δυναμικό. Υποστηρίζουμε την υιοθέτηση της Δευκής Βούγκτου για την άμυνα με βάση την παγκόσμια στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την κοινή εξωτερική πολιτική, επανεξετάζοντας ε, την κατάσταση και 7. την ανάγκη να εξασφαλίσουμε την στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Έχω και 66 τροπολογίες πέρα από τις 7 αυτές προτάσεις και θα τις εξετάσουμε τις επόμενες μέρες αυτές τις τροπολογίες, αλλά πιστεύω θα βρούμε καλές συμβαστικές ε, προτάσεις μεταξύ των πολιτικών ομάδων και θα κινηθούμε και προς τη γραμμή που μας ανέπτυξε και ο εισηγητής. Ευχαριστώ κύριε Μακάλιστερ. Και τώρα περνάμε στις συνεισφορές των σχεδόν συγητών. Ο κύριος Μάικλ Γκάλερ από το ΕΛΚΑ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση. Υπάρχει μια αρκετά ευρεία συνένεση, όχι μόνο στο Κοινοβούλιο, αλλά και στο Συμβούλιο. Υπάρχουν άτομα τα οποία ενδιαφέρονται. Ο Γερμανός Υπουργός Άμυνας είπε στο Βίλνιους όταν έγινε μια συνάντηση πριν από δύο εβδομάδες ότι πραγματικά ενδιαφερόμαστε. Πιστεύω πως είναι καιρός να προχωρήσουμε προς μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση. Ήταν η Ούρσουλα Φόντερ Λάιν που έκανε αυτή την παράθεση. Καλωσορίζω επίσης την έκθεση του συναδέλφου μας ΠΑΤ. Είναι και ώρα, νομίζω, να περάσουμε σε μια νέα φάση των συζητήσεων και να ενεργοποιήσουμε τις διατάξεις της συνθήκη προς αυτή την κατεύθυνση, με αυτό το σκοπό. Ως ε, μέλος του ΕΛΚ καλωσορίζω την έκθεση του συναδέλφου και το ΕΛΚ συνολικά καλωσορίζει την έκθεση γιατί δίνει τη δυνατότητα να εκφράσουμε τις απόψεις του Κοινοβουλίου για τη συνέχεια που θα πρέπει να δοθεί στην παγκόσμια στρατηγική στα πλαίσια της ασφάλειας και της άμυνας. Θα θέλαμε να υπάρξει ένα έγγραφο υπομορφή λευκής βίβλου για να δούμε πώς θα προχωρήσουμε προς αυτή την αμυντική ένωση. Ε, στη φάση της, του σχεδίου εφαρμογής ε, αυτό που προβλέπουμε δηλαδή σε αυτή τη φάση, το σχέδιο αυτό εφαρμογής, εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι αρκετό. Θέλουμε λοιπόν κάτι παραπάνω, ένα κείμενο follow-up. Οι απόψεις μας ε, θα παρουσιαστούν και από την κυρία Μογκερίνη αύριο στη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας στην... Θα τις παρουσιάσουμε μάλλον στην κυρία Μογκερίνη ε, στη συνάντηση στην Πρατισλάβα. Η έκθεση κινείται προς σωστή κατεύθυνση και γενικά συνάδει με τις ε, θέσεις μας. Θα ήθελα να προσθέσω ίσως λίγα στοιχεία. Καταρχάς, καλωσορίζουμε την υποστήριξη της Γερμανίας, Γαλλίας, ε, Ιταλίας, ε, ε, Ολλανδίας και κάποιων κεντροευρωπαϊκών χωρών για μεγαλύτερη ολοκλήρωση σε αμυντικά θέματα και ακούσαμε και πολύ καλές δηλώσεις και πολύ ενθαρρυντικές προς αυτήν την κατεύθυνση. Αυτές οι ανακοινώσεις μου δίνουν αισιοδοξία. Και η διαδικασία της Λευκής Βίβλου θα οδηγήσει σε αυτή την αμυντική ένωση. Ζητήσαμε μια αμυντική αναθεώρηση ούτω ώστε να κάνουμε μια αποτίμηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Καταρχάς, να δούμε τι έχουμε πριν αρχίσουμε να σχεδιάζουμε τα επόμενα βήματα. Εν συνεχεία, θα πρέπει να έχουμε αυτόν τον κοινό αμυντικό σχεδιασμό, να δούμε τι ε, ευρωπαϊκό, ευρωπαϊκό δυναμικό έχουμε με βάση το άρθρο 42 της συνθήκης. Επίσης, μια αναθεώρηση της οργάνωσης και των διαδικασιών και των δραστηριοτήτων ε, τη Ευρωπαϊκή Αμυντική ε, Υπηρεσία του οργανισμού, ούτω ώστε η ΕΝΤΑ, ο Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα, να είναι κατάλληλο για τα μελλοντικά καθήκοντα. Για δύο λόγου. Καταρχά τα τελευταία χρόνια είδαμε ότι υπάρχει ένα δημοσιονομικό αδιέξοδο. Τα κράτη-μέλη έχουν βάλει ε, ένα φραγμό για την αύξηση του προπολογισμού, ειδικά τα κράτη τα οποία είναι προ την έξοδο. Δεν θα πρέπει να συνεχίσουν να μπλοκάρουν τι δραστηριότητε τη ΕΝΤΑ, αλλά νομίζω ότι Υπάρχει και ένα πρόγραμμα για αμυντική έρευνα ε, από την επόμενη περίοδο, δηλαδή από το 2021 και μετά, και αυτό θα πρέπει να γίνει. Μιλάμε για 3,5 περίπου δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, ο σημερινό ευρωπαϊκό άμυνα με τη σημερινή του μορφή, με το μέγεθο που έχει κτλ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να διαχειριστεί ένα τέτοιο προπολογισμό και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνει μια αναφορά στην ανάγκη να αναθεωρήσουμε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνα, ακριβώ και για αυτόν τον λόγο. Για τα λεφτά. Ναι, σίγουρα θα πρέπει να αυξήσουμε την ε, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για την αμυντική άμυνα ε, μέσω αυτή τη προπαρασκευαστικής δράση και με βάση το πιλωτικό σχέδιο που είχε ετοιμάσει το Κοινοβούλιο στα πλαίσια του προπολογισμού του 2015 και του 2016. Καταλαβαίνουμε βεβαίω τι ανησυχίε του εισηγητή για τον προπολογισμό του 2017, ε, που θεωρεί ότι η αμυντική έρευνα ε, έχει προβλήματα. Ο, και μιλάω για το γενικό ε, εισηγητή του προπολογισμού. Υπάρχει μια ευρεία ε, συνένεση στο Κοινοβούλιο ότι αυτή η προπασκευαστική δράση που προτείνει η Κομισιόν θα πρέπει να γίνει. Η ασφάλεια και η άμυνα είναι ψηλά στην ατζέντα της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, να σας παραπέμψω και στα όσα είπε το Συμβούλιο και στις δημοσιονομικές δεσμεύσεις οι οποίες θα πρέπει να παρακολουθούν και να εντάσσονται μέσα στα πλαίσια αυτών των νέων προτεραιοτήτων για την άμυνα. Από τους σοσιαλιστές, ο κύριος Τονίνο Πικούλα. Thank you. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον συνάδελφο για την έκθεσή του. Όπως υπόθηκε και πιο πριν, είναι καιρός για αυτή την έκθεση. Πριν από μια εβδομάδα οι ηγέτες της Γαλλίας, της Ιταλίας και της Γερμανίας έστειλαν ένα σαφές μήνυμα πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να αυξήσει έντονα τη συνεργασία της στην άμυνα και στις πληροφορίες. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση προκαλούν μια αλλαγή της τάσης προς την κατεύθυνση μιας Ευρωπαϊκής Αμυντικής Ένωσης. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε την πολιτική, την πολιτική στιγμή αυτή για να κάνουμε συγκεκριμένα βήματα προς την περαιτέρω ολοκλήρωση της πολιτικής άμυνας. Μόνο τέσσερα κράτη-μέλη, στην πραγματικότητα μόνο τρία, επειδή ένα εξ αυτών είναι το Ηνωμένο Βασίλειο, επιτυγχάνουν, πληρούν τον στόχο του ΝΑΤΟ να επενδύουν 2% του ΑΕΠ του στην άμυνα. Πρόκειται για μια πρόκληση για την άμυνα. Γι' αυτό και υποστηρίζω την γραμμή του εισηγητή όσον αφορά τα έξοδα για την άμυνα και την σχέση με τα ευρωπαϊκά ταμεία η επένδυση στην άμυνα και ιδίω στην έρευνα μπορεί να αποτελέσει μια μεγάλη ευκαιρία για οικονομική ανάπτυξη. Επίσης υποστηρίζω την πρόταση του εισηγητή για τη Λευκή Βίβλο ασφάλεια και Άμυνας. Περαιτέρω πιστεύω πως πρέπει να πάμε πιο μακριά από το στρατηγικό πλαίσιο. Στην επίκυρη κατάσταση ασφαλεία οι πολιτικές ασφάλειας και άμυνας θα πρέπει, δεν θα πρέπει να είναι ο πιο αδύναμος σύνδεσμος στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να δημιουργήσει την ταυτότητά της στον 21ο αιώνα μέσω ασφάλειας και άμυνας και θα αξιολογηθεί με βάση το αν θα μπορέσει να εγκαθιδρύσει ένα επαρκές σύστημα προστασίας των πολιτών της. Εάν αποτύχουμε να προσφέρουμε την ασφάλεια στους πολίτες μας, τότε αυτοί θα αποξενωθούν. Ολοκληρώνοντας αυτό το σχέδιο έκθεσης δίνει μια καλή βάση για συζήτηση επί της οποίας μπορούμε να επικοδομήσουμε και προσμένουμε χαρά την μελλοντική μας συνεργασία. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Εκ μέρους του ECR, Τζεφρή Βανόρτεν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Όπως γνωρίζετε, έχω κάποιες θεμελιώδεις δυσκολίες με αυτές τις έννοιες για την όλη συζήτηση αυτή για την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση η οποία χαρακτηρίζεται από μια έλλειψη ειλικρίνειας. Η επιχειρηματολογία ακούγεται εύλογη ιδίως για τον παρατηρητή εκ των έξω θα πρέπει να αναγνωρίσουμε πως επί 70 χρόνια τα ευρωπαϊκά έθνη αφενός και ο μεγάλος σύμμαχός τους, οι Ηνωμένε Πολιτείε, αγωνίστηκαν για να βρουν έναν τρόπο για να συνεισφέρουν οι Ευρωπαίοι περισσότερο στην, στην υπεράσπιση των ελευθεριών τους. Οι Βρετανοί και οι Αμερικανοί είχαν μια πραγματιστική αντίληψη για την άμυνα αλλά για άλλα έθνη. Μια νέα ιδεολογική, ένα ιδεολογικό συστατικό ενσωματώθηκε στην προσέγγιση. Αυτό το ευρωπαϊκό κράτος το οποίο θα έχει δικές του ε, ένοπλες δυνάμεις και δεδομένης της σημασίας των ένοπλων δυνάμεων ως μέσο άσκησης κυριαρχικών δικαιωμάτων μιας Ευρώπης με κεντροποιημένο προϋπολογισμό θα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα πολιτικά βήματα προς την δημιουργία ενός ευρωπαϊκού κράτους. Περί αυτού πρόκειται. αν σκεφτούμε τις αρχές της δεκαετίας του 50, της τότε ιδέας της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Άμυνας. Αυτό φυσικά ήταν μια πρόταση εν της σοβιετικής απειλής, να βρεθεί ένας τρόπος να δημιουργηθούν στρατιωτικές ικανότητες στη Γερμανία χωρίς να επανεξοπλιστεί η Γερμανία. Περί αυτού επρόκειτο τότε. Έκτοτε η έμφαση μετατοπίστηκε. Υπάρχει μια διαφορά μεταξύ αυτών που θέλουν να ολοκληρώσουν την Ευρώπη σε πολιτικό επίπεδο και σε αυτόν που αποζητούν περισσότερη στρατιωτική ισχύ. Και τα δύο δεν είναι κατά ανάγκη συμβατά. Και πιστεύω πως πρόκειται για μια ανηλικρινή κίνηση να λέγεται στους Αμερικανούς πως οι αμυντικές φιλοδοξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι προς συμφέρον της Αμερικής. Γνωρίζουμε την συζήτηση για την κατανομή των βαρών η οποία συνεχίζεται μετά από 70 χρόνια. Αυτό δεν είναι η απάντηση. Θα έχει το ακριβώς αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που θέλουν σε τελική ανάλυση οι μεγάλοι Αμερικανοί σύμμαχοί μας. Δεν θα δημιουργηθούν έτσι περισσότερες στρατιωτικές ικανότητες, αλλά διέρεση, πόλωση με τους Ευρωπαίους από τη μία πλευρά και τους Αμερικανούς από την άλλη. Θα δημιουργηθεί έτσι ένας εταίρος σε απόσταση που δεν θα έχει αξιοπιστία. Μου λέτε ειλικρινά πως η Μόσχα, για παράδειγμα, θα ανησυχεί πράγματι για κάποια δυνητική Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση ή ανησυχεί περισσότερο η Μόσχα για το ΝΑΤΟ όπως είναι με συμμετοχή των Ηνωμένων Πολιτειών πού θα βρίσκεται η αξιοπιστία σε αυτή την Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση. Επίσης θα ήθελα να τονίσω πως δεν υπάρχει καμία ανάγκη να εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Ένωση σε οποιοδήποτε από αυτά τα ζητήματα. Ήδη έχουμε αμυντική βιομηχανική συνεργασία χωρίς την εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ήδη υπάρχουν πολυεθνικές στρατιωτικές ομάδες, μονάδες, οι οποίες υπάρχουν εδώ και δεκαετίες χωρίς να έχει εμπλακεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό δεν πρόκειται για ανακάλυψη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει εδώ και δεκαετίες. Και επίσης υπάρχουν αμυντικές υποδομές χωρίς εμπλοκή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό που βλέπουμε σήμερα στην έκθεση αυτή και σε παρόμοιες εκθέσεις που καταθέτονται αυτή τη στιγμή είναι αυτή η όθηση προς την κοινοτικοποίηση της άμυνας η ευρωπαϊκή κοινότητα δεν έχει κανένα ρόλο στην άμυνα ή δεν θα πρέπει να έχει. Αυτό είναι ένα ζήτημα που αφορά τα έθνη. Αλλά αυτή τη μετατόπιση θέλουν να δουν οι άνθρωποι. Μιλούμε για την εταιρική σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Για τι πράγμα μιλάμε. Ας πούμε την αλήθεια. Είναι, μιλούμε για έθνη. Και τα ίδια έθνη, εκτός από ένα που αποκλείεται, στο ένα μοντέλο αποκλείονται οι Ηνωμένε Πολιτείε, στο άλλο συμμετέχουν. Φυσικά και θα μπορούσε να υπάρξει μια χρήσιμη εταιρική σχέση μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ. Εάν η Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεντρωνόταν σε αυτό που θα μπορούσε να κάνει επιπρόσθετα, εκεί που θα μπορούσε να προσθέσει αξία. Και κυρίες και κύριοι, αυτό δεν είναι στο στρατιωτικό τομέα, αλλά στον πολιτικό. Ίσως, αν χρησιμοποιούσε τους πόρους της διαφορετικά και πιο εύλογα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει κάτι να προσθέσει όσον αφορά την διαχείριση κρίσεων και θα μπορούσε να ασχοληθεί με την επίλυση συγκρούσεων, με την αποκατάσταση και με όλα αυτά τα ζητήματα, ναι, την ανθρωπιστική βοήθεια. Υπάρχουν πολλά που θα μπορούσε να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση συμπληρωματικά προς τον ΝΑΤΟ. Αλλά αυτό που δεν χρειάζεται να κάνει είναι να δημιουργήσει τη δική του ξεχωριστή αυτόνομη στρατιωτική δομή. Ιδίω σε μια εποχή στην οποία οι αμυντικοί πόροι είναι περιορισμένοι και φυσικά βλέπουμε πολλές χώρες που πιστεύουν ότι θα λάβουν φτηνή άμυνα, ότι θα υπάρξει μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση η οποία θα αναλάβει την ευθύνη και θα φέρει το βάρος αντί τα ίδια τα κράτη να κάνουν περισσότερα. Ας σας θυμίσω κάτι κυρίες και κύριοι. Όταν το Ηνωμένο Βασίλειο αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μειωθεί δραστικά. Την ίδια στιγμή ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός θα μειωθεί σημαντικά. Πολλοί από ό,τι φαίνεται δεν αντιλαμβάνονται πως το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εισφορέας στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εδώ πολλοί πιστεύουν ότι η Γερμανία πληρώνει για τα πάντα. Κι όμως δεν είναι έτσι. Πληρώνεται πολύ, αλλά εξίσου το Ηνωμένο Βασίλειο. Και αυτό θα σταματήσει. Και είναι κάτι άλλο για το οποίο δεν μιλούν οι άνθρωποι αυτή τη στιγμή ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι σημαντικά πιο μικρός. Κυρίες και κύριοι, δεδομένων των απειλών που αντιμετωπίζουμε όλοι και των απειλών για την, τις δυτικές δημοκρατίες, οι οποίες είναι ίδιες στη Βαρσοβία, στο Βερολίνο, στο Παρίσι, στην Ουάσιγκτον. Χρειαζόμαστε αλληλεγγύη μεταξύ των δυτικών συμμάχων. Χρειάζεται να κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρήση των, ε, της δομής η οποία μας χρησιμεύσε τόσο επί δεκαετίες, η οποία είναι το ΝΑΤΟ. Και μην αποπλανηθείτε τώρα από τους μάγους αυτούς που σας κοροϊδεύουν, υποστηρίζοντας ότι μια Ευρωπαϊκή Αμυντική Ένωση είναι η απάντηση για όλα τα προβλήματά μας. Το αντίθετο ισχύει. Πρόκειται για ένα επικίνδυνο βήμα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστούμε, ε, κύριος Πάσκου. Ευχαριστώ. Και πάλι έχουμε επιστρέψει στο μηδέν. Στη, από εκεί που ξεκινήσαμε, τα έχουμε ξανασυζητήσει με τον Τζέφρι, λέει ότι η Μόσχα δεν μπορεί να μας πάρει στα σοβαρά στον αμυντικό τομέα. Εγώ θα έλεγα ότι η τακτική της Μόσχας είναι το Δίρι και Βασίλευε. Και το ότι οι Ευρωπαίοι βρίσκουν έναν τρόπο για να ε, εντατικοποιήσουν τη συνεργασία τους στέλνει το σωστό μήνυμα στους Ρώσους ότι αυτή η τακτική τους εμάς δεν θα περάσει. Ειδικά για τα θέματα ασφάλειας και άμυνας. Νομίζω Πώς μπορείς, ε, Τζέφρι, να εξακολουθείς να επιμένεις στην άποψή σου. Και εγώ το ίδιο. Και η ζωή θα, θα αποδείξει ποιος είχε δίκαιο στο τέλος. Δε, πρώτον. Δεύτερον, είπες ότι θα είναι περιορισμένος ο προπολογισμό. Μα το Ηνωμένο Βασίλειο τα τελευταία χρόνια μου μας εκπαίδευσε ε, να έχουμε περιορισμένα κονδύλια, γιατί εκείνη ε, εσείς επιμένατε ότι θα αποχωρήσετε άμα αυξηθούν υπερβολικά τα κονδύλια. Θα μας έλεγε ο Κάμερον. Οπότε μην ανησυχείς, συνηθισμένα τα βουνά στα χιόνια. Θα τα καταφέρουμε και με λίγα λεφτά. Νομίζω ότι με τους Αμερικανούς εδώ, αυτό είναι το παιχνίδι και θα το συζητήσουμε σήμερα, θα, θα, θα έχουμε το debate σήμερα των Αμερικανών και μάλλον θα ξεκαθαρίσει η εικόνα μετά. πρέπει να ξέρεις ότι εκείνοι θα αποφασίσουν ε, ανάλογα με το ποιος θα υποψήφιος θα επικρατήσει. Και θα πρέπει να προφυλαχθούμε κι εμείς ε, ε, για αυτό το ενδεχόμενο ως Ευρωπαϊκή Ένωση. Επίσης δεν είναι πάντοτε ευπρόσδεκτη σημαία του ΝΑΤΟ. Καμιά φορά, όπως πολύ καλά ξέρουν όλοι, χρειάζεται μια διαφορετική σημαία. Εσύ κυρίως τα ξέρεις αυτά. Και γι' αυτό θα πρέπει να λειτουργήσει αυτό ως κίνητρο. Πάμε να πιούμε ένα, μια μπύρα στην ε, Ιρλανδέζικη Παμπ και να μην μαλώνουμε. Και ε, όποιος ζήσει αρκετά θα δει ε, ποιος από τους δύο είχε δίκιο. Ευχαριστώ. Μπαρμπότζο Παραγιούρκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ, Φρέδρε. Χαίρομαι που συζητούμε αυτό το θέμα. Έχουμε μια σοβαρή κρίση να αντιμετωπίσουμε και θα πρέπει να αντλήσουμε τα εξή συμπεράσματα. Αυξάνονται οι εθνικέ εθνικές δαπάνε. δαπάνες και ε, δεύτερον ε, θα πρέπει να δείξουμε αλληλεγγύη και κυρίως αλληλεγγύη στα σύνορα είναι σημαντικό να μιλήσουμε για τα ζητήματα αυτά. Στο σημείο 11 υπάρχει, υπάρχει μια έκκληση για αύξηση εξόδων. Στο 9 υπάρχει η σύσταση να ενταθεί η συμβατότητα των προσπάθειων της συμβατότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ και στο 16 υπάρχει μια έκκληση αλληλεγγύης στα ευρωπαϊκά σύνορα, εκεί αφορά τα βαλτικά κράτη. Αλλά εκεί δεν έχουμε παραλέξεις επειδή η αύξηση των εξόδων αυτό δεν μπορεί παρά να αποτελεί ε, έκκληση ή μάλλον σύσταση. Η χώρα μου ανήκει στις λίγες οι οποίες πληρούν πλήρως τις υποχρεώσεις αυτές. Δεύτερον, περισσότερη πολιτική αλληλεγγύη πρόκειται για ορισμένες δεσμεύσεις. Θέλουμε να δημιουργήσουμε συγκεκριμένες πολιτικές δομές μόνο με ανθρωπιστικά καθήκοντα και όχι με αμυντικά. Και τρίτον, η συνοριακή αλληλεγγύη. Η προσάρτηση της Κρυμαίας έχει περάσει πολύ καιρός από τότε, αλλά πραγματικές αντιδράσεις δεν υπήρξαν σχεδόν καθόλου. Όσον το πιο αξιόπιστο στοιχείο της έκθεσης αυτής είναι η συνθήκη της Λισαβόνας. Αλλά η συνθήκη της Λισαβόνας οδήγησε στο Brexit. Οπότε το ερώτημα είναι κατά πόσο να αξίζει το κόπο να συνεχίσουμε σε αυτό το δρόμο ή κατά πόσο θα έχει νόημα στην αρχή να θεσπίσουμε μια κοινή πολιτική, να υλοποιήσουμε συγκεκριμένους στόχους. Παραδείγματος χάρη η καθολικοποίηση του στόχου των 2% του ΑΕΠ για αμυντικά έξοδα και παραδείγματο χάρη επίση στρατιωτική παρουσία και όχι μόνο η ζήτηση αμερικανική βοήθεια. Εάν εμεί βοηθήσουμε του εαυτού μα, τότε δεν θα χρειάζεται να ζητούμε μόνο τη βοήθεια των ΗΠΑ. Και αυτή χρειαζόμαστε μια πραγματική αλληλεγγύη εκεί όπου οι κίνδυνοι είναι μεγαλύτεροι. Και δεν σκέφτομαι μόνο την κεντρική και την ανατολική Ευρώπη. Αλλά αυτό ισχύει επίση για τον χώρο τη Μεσογείου. Α σκεφτούμε πω πριν από 1,5 χρόνο είχαμε στρατιωτικέ δράσεις ενάντια στη μαφία των διακινητών. Αλλά αυτές περιορίστηκαν μόνο σε ανθρωπιστικά μέτρα, τα οποία ήταν πολύ χρήσιμα, αλλά αποκλίνει πολύ από αυτό που συμφωνήθηκε πέρυσι τον Απρίλιο. Θα επαναλάβω, αξίζει να θέσουμε επαμφιβόλο το δρόμο της Λισαβόνας και να σκεφτούμε με διαφορετικό τρόπο για την αλληλεγγύη, με την ελπίδα πως με την αλληλοβοήθεια θα επιτύχουμε καλύτερα αποτελέσματα και θα ήταν χύμπερα να νομίσουμε ότι οι νέοι θεσμοί λύνουν τα προβλήματα από μόνοι τους. Αυτό δεν έχει λύσει μέχρι στιγμής κανένα πρόβλημα. Ευχαριστώ. Θα γίνει και δεύτερος γύρος. Ο κύριος ε, Γκάλε ε, θέλει να ξαναπάρει το λόγο. Θα είμαι όμως εγώ, αν μου το επιτρέπετε, η τελευταία μιλήτρια του πρώτου γύρου. Απευθύνω προς τους εισηγητές. Πώς τοποθετήσετε σε σχέση με, ε, με μια ενιαία αντίληψη των κινδύνων Και για τους σκοπούς της συζήτησης θέλω να πω ότι εκπροσωπούμε και την Κεντρική και την Ανατολική Ευρώπη και αν υπάρχει ξεκάθαρη βούληση ε, σε εμπόλεμες ζώνες στον Νότο να σταλούν μάχημες ομάδες ε, στα πλαίσια της πολιτικής ε, ε, τότε θα ξαφνιαστώ. Εγώ δεν έχω δει, ας πούμε, πολιτική βούληση σε σχέση με το αίτημα της Ουκρανίας ε, να υπάρξει αποστολή ε, και επαϊκή. Διαβλέπετε εσείς ε, δυνατότητα να υπάρξει κοινή προσέγγιση για τις κοινέ απειλές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και δεύτερον, απηχώντας αυτά που είπανε η κύριοι Γκάλα και Βανόρντεν για το ρόλο του Ηνωμένου Βασιλείου ε, και τη συμβολή του ε, στη χρηματοδότηση, δηλαδή στον προϋπολογισμό. Όταν μιλάμε για τις μελλοντικές ευρωπαϊκές δαπάνες ε, στον αμυντικό τομέα, Δεν πρέπει να ξεχνάμε, ήταν πάγια θέση του Ηνωμένου Βασιλείου. να διαθέτει ένα μεγάλο κομμάτι του εθνικού προϋπολογισμού για, για τη χρηματοδότηση αμυντικής ικανότητας. Σε κάποια κράτη-μέλη υπάρχουν πραγματικές αμυντικές ικανότητες και αυτό μπορεί να προσδώσει μια προστιθέμενη αξία στις προσπάθειές μας. Εσείς ε, πώς τοποθετήσετε, πώς μπορούμε να ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα, πώς ενδεχομένως μπορούμε να εξασφαλίσουμε τη συμμετοχή ε, του Ηνωμένου Βασιλείου, τη συνεργασία του Ηνωμένου Βασιλείου με εμάς ε, σε ένα θεσμικό πλαίσιο. Τώρα, θα δώσω το λόγο ε, στον κύριο Γκάλλο δεύτερη φορά και μετά στον κύριο Απάτη, γιατί ξέρω ότι βιάζεται. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Για να το καταστήσω σαφές, η πολιτική ομάδα του ΕΛΚ θεωρεί τις δραστηριότητες και τη μετεξέλιξη της ΚΠΑ ως ενδυνάμωση του ευρωπαϊκού πυλώνα του ΝΑΤΟ. Αυτό δεν, είναι, δεν σημαίνει ότι θέλουμε να βγούμε από το ΝΑΤΟ ή θέλουμε να το κάνουμε έναν οργανισμό δεύτερης κατηγορίας του αντίον. Το ζητούμενο είναι να συγκεντρώσουμε τις δυνάμεις μας κατά τέτοιον τρόπο ώστε να μπορούμε να έχουμε να επιτύχουμε μια πιο δυνατή συνεισφορά στα πλαίσια του ΝΑΤΟ και η καταγγελία από τις Ηνωμένε Πολιτείε, ότι είμαστε free riders στο ζήτημα της άμυνας πιστεύω πως μπορούμε να απαντήσουμε στην κατηγορία αυτή. Έχουμε δυνατότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο, παραδείγματος χαρί στην εσωτερική αγορά, επειδή θεωρητικά έχουμε την ενιαία αγορά αμυντικών προϊόντων. Θεωρητικά αυτό ισχύει ήδη, αλλά τα κράτη-μέλη αποχωρούν συνεχώς. Πιστεύω ότι τα χρήματα που έχουμε μπορούμε να τα ξοδέψουμε καλύτερα. Και πιστεύω πως στην πραγματικότητα με καλύτερο κοινό σχεδιασμό και καλύτερες κοινέ προμήθειες μπορούμε να εξοικονομήσουμε πολλά χρήματα και να αυξήσουμε την διαλειτουργικότητα. Εάν κάναμε πολύ περισσότερα από κοινού. Επειδή όταν είμαστε σε μία αποστολή, κατά 99% είμαστε στους ίδιους τόπους σε αποστολή. Και όταν είμαστε στο ίδιο, στον ίδιο τόπο, χρειαζόμαστε τα ίδια οπλικά συστήματα και τις ίδιες ικανότητες. Γι' αυτό και δεν βλέπουμε κάποια αντίφαση ως προς αυτό. Και κυρίως ο συνάδελφος Μπάσπουτ το έθεσε σωστά, η σημαία του ΝΑΤΟ δεν είναι παντού εξίσου καλοδεχούμενη, Αυτή είναι μία εκδοχή. Αλλά ίσω υπάρχει και ο ένα ή άλλος εταίρο του ΝΑΤΟ που δεν θέλει η Ευρωπαϊκή Ένωση να ενεργοποιηθεί ω Ένωση. Και πριν από το πραξικόπημα, αλλά και τώρα. Χρησιμοποιώ το παραδείγμα της Τουρκίας. Τι θα κάνουμε εάν χρειαστεί, αν θελήσουμε να χρησιμοποιήσουμε πόρους του ΝΑΤΟ ως Ευρωπαϊκή Ένωση, αν πούμε ότι θα πάμε στη Λιβύη και ο κύριος Ερντογάν δεν το θεωρεί σωστό. Τότε θα ασκήσει βέτο, ακυρώνοντας οτιδήποτε θα μπορούσε να γίνει στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, που οι αποφάσεις λαμβάνονται επίσης με αυτονομία. Γι' αυτό και χρειαζόμαστε μια στρατηγική αυτονομία για αποστολές, τις οποίες θέλουμε να προβούμε, προς το δικό μας κοινό ευρωπαϊκό συμφέρον. Και γι' αυτό το λόγο πιστεύω ότι είναι σωστό να πάρουμε το δρόμο αυτό προς την αμυντική ένωση. Και όσον αφορά την κοινή πρόσληψη της ασφάλειας, παρέπεμψα ήδη στη δήλωση της Υπουργού Αμήνισμου. η δήλωση έγινε στο Βίλνιους. Ίσως θα έπρεπε να το πει στη Ρώμη. Θα ήταν ακόμα καλύτερο. Επειδή ίσως αναφορικά με την Ανατολή, στη Ρώμη, η ευαισθησία είναι διαφορετική από ό,τι είναι ούτως ή άλλως στο Βίλνιος ή στο Βερολίνο. Ευχαριστώ. Μάλιστα. Ο κύριος Φανόρτεν ξαναζήτησε το λόγο. Πολύ σύντομα. Δεν θα να τη συζήτηση. Κοιτάξτε το, εάν έχετε αυτόνομη διαδικασία λήψη αποφάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση για τα αμυντικά θέματα. Αν έχετε χωριστές ευρωπαϊκές δομές, πώς θα ενισχύσουμε με αυτόν τον τρόπο την, πώς ενισχύει με αυτόν τον τρόπο την αλληλεγγύη. Αυτό αντίθετα δημιουργεί διχασμούς, διαιρέσεις, ρήγματα. Φυσικά και το κάνει. Αν έχουμε μια κρίση, θα πρέπει κανονικά μαζί με τους Καναδούς, τους Αμερικανούς λοιπά να καθίσουμε γύρω από ένα τραπέζι για να αντιμετωπίσουμε με τον καλύτερο τρόπο αυτή την κρίση. Μπορεί σε ορισμένε περιπτώσει οι Ευρωπαίοι να έχουν τον ηγετικό ρόλο. Αλλά Μάικλ, εσύ μίλησε για τη Λιβύη. Φυσικά, επειδή είσαι Γερμανό, είναι ενδιαφέρον το, το ότι μιλησε για τη Λιβύη, γιατί οι Γερμανοί αρνήθηκαν να συμμετάσχουν στις επιχειρήσεις για, στη Λιβύη. Α, μιλάς ως Ευρωπαίος τώρα, έτσι, ως μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος πάντων, κακό παράδειγμα διάλεξες. Και όμως εγώ θεωρώ ότι είναι καλό παράδειγμα η Λιβύη. Γιατί αν η Ευρωπαϊκή Ένωση θα, θα ήθελε να εμπλακεί σε κάποιες επιχειρήσεις, ποιος θα υποστηρίξει τους Ευρωπαίους. Ποιος θα τους ε, βοηθήσει οικονομικά όταν ε, αντιμετωπίσουν ε, δυσκολίες. Ποια δύναμη θα έρθει να τους βοηθήσει να τους διασώσει. Εκτός μικροφώνου παρεμβάσεις. Δεν είναι σοβαρές απόψεις αυτές, ενώ θα έπρεπε να είμαστε σοβαροί. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα πιο σοβαρό από τις ε, προκλήσεις ασφάλειας που αντιμετωπίζουμε. Και εσείς συνέχεια μιλάτε για το πώς θα πάει μπροστά η Ευρωπαϊκή Ένωση, πώς θα παίξει τον πολιτικό της ρόλο κτλ. Σας παρακαλώ, ας πούμε τα πράγματα με το όνομά έτσι, και ας μην κρυβόμαστε πίσω από τα λόγια. Συγγνώμη. Νομίζω ότι εγώ κανονίζω τη συζήτηση. Θέλετε να δώσετε κάποια απάντηση. Ο κύριος ε, Ούρμας Πατ. Ε, σας ευχαριστώ για τις παρατηρήσεις, τα σχόλια και τις προτάσεις. Ε, συμφωνώ. Φυσικά υπάρχουν αμυντικά ευρωπαϊκά θέματα τα οποία θα πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε ως τέτοια. Ε, να λάβουμε υπόψη μας τις διαφορές, αλλά υπάρχει και το άρθρο 42 στη συνθήκη, που είναι κενό περιεχομένο. Το είδαμε πριν από κάνα χρόνο και μετά τις ε, επιθέσεις στο Παρίσι, που ζήτησε η Γαλλία, ας πούμε, συγκεκριμένη βοήθεια από άλλες ευρωπαϊκές χώρες και ξέρουμε πολύ καλά Ποια ήταν η απάντηση, η απόκριση των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών σε αυτό το αίτημα. Επίση, η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωση για θέματα άμυνα επισύρει πολλέ κριτικέ και από την πλευρά του ΝΑΤΟ. Ότι δεν υπάρχει αρκετή υποστήριξη, δεν δείχνει εταιρικότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτέ οι κριτικέ ακούγονται εδώ και χρόνια. Και υπάρχουν και πολλά πρακτικά πράγματα τα οποία μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση πολύ καλύτερα. Πιστεύω πραγματικά ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι έτοιμη να κάνει πολύ περισσότερα εάν εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχουν πολύ πιο συγκεκριμένοι κανονισμοί, σας αρέσει ή δεν σας αρέσει, έτσι είναι τα πράγματα. Πολλά πράγματα γίνονται και στα κρατη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση όταν υπάρχουν σαφείς κανονισμοί και γενικά κανόνες. Όταν έκανα τις αρχικές μου παρατηρήσεις, είπα ότι το ΝΑΤΟ αποφασίζει να στείλει περισσότερα στρατεύματα τώρα σε ορισμένε ανατολικέ Ευρω... χώρε τη ε, της Ανατολικής Ευρώπης δηλαδή. Να ένα πράγμα που μπορεί να κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεισφέρει στην υποδομή, στην επιμελητία ε, για να βοηθήσει ας πούμε ε, με στρατώνες ας πούμε αυτά τα στρατεύματα. Υπάρχουν πάρα πολλά θέματα τα οποία μπορεί να βοηθηθούν, στα οποία η Ευρωπαϊκή συνεργασία με την νατοϊκή συνεργασία μπορεί να τα προωθήσει. Επίσης, γεγονός είναι ότι η πλειοψηφία των χωρών του ΝΑΤΟ είναι μέλη ταυτόχρονα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν όμως και ευρωπαϊκές χώρες που δεν είναι μέλη του ΝΑΤΟ. Κάποιες σκανδιναβικές, Αυστρία, Ιρλανδία κλπ. Ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να είναι, λοιπόν, όλες αυτές οι χώρες να εμπλακούν. Και αυτό που ανησυχεί το Ηνωμένο Βασίλειο τελικά. Να σας πω, εγώ υποκειμενικά μιλάω, έτσι. Αυτό συνδέει το Ηνωμένο Βασίλειο με την υπόλοιπη Ευρώπη. Αν είναι κάτι που τη συνδέει πιο έντονα από οτιδήποτε άλλο, είναι τα αμυντικά θέματα. Τώρα, για τα συγκεκριμένα δημοσιονομικά θέματα, τον προπολογισμό κτλ. Κανένα δεν ξέρει. Θα δούμε στι διαπραγματεύσει τι θα γίνει. Είναι ξεκάθαρο όμω ότι δεν έχει κανένα νόημα να λέμε ότι η Ευρώπη θα αναπτύξει τη δική της ασφάλεια και άμυνα μόνη της, χωρίς να εμπλακούν και σημαντικέ ευρωπαϊκέ χώρε οι οποίε δεν είναι μέλη τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι ρεαλιστικό, το ξέρουμε. Επομένω, μία συνεργασία με το Ηνωμένο Βασίλειο είναι απολύτω εκ των ονουκάνων. Η δεύτερη εξέταση της έκθεσης θα γίνει τον Οκτώβριο στις 12 του μηνός. 12 και 13 η συνεδρίαση. Και από ό,τι ξέρω, οι σκιώδεις συζητητές θα συναντηθούν αύριο. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πατ. Και πάμε στο επόμενο σημείο, που είναι η ενημέρωση. για την αποστολή της έντες στο Μαλί. έγινε από τις 18 στις 21 Ιουλίου, το 16 φυσικά, το πρόγραμμα το ετοίμασε ο συνήθως η γραμματεία, ήταν πολύ πλούσιο. Καταρχάς, καταφέραμε να συναντήσουμε τους διοικητές και μέλη του επιτελείου της ε, Ευρωπαϊκής Αποστολής στο Μαλί. Του συναντήσαμε και στην πρωτεύουσα, του Παμάκο. και στα γραφεία και στους χώρους εκγύμνασης μιλήσαμε με προσώπους των προέδρων των, επιτροπών, των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Άμυνας, μιλήσαμε ε, με τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Δυστυχώς, λόγω μιας μεγάλης τρομοκρατικής επίθεσης που έγινε κατά τη διάρκεια της παραμονής μας, κοντά στα σύνορα με τη Μαυριτανία, εναντίον στρατιωτικών δυνάμεων του Μαλή, δεν μπορέσαμε να, να συναντήσουμε μέλη της κυβέρνησης και συνεργάτες του Προέδρου. Όμως, θεωρούμε ότι η αποστολή αυτή ήταν πολύ επωφελής. Η αξιολόγηση των επιχειρήσεων και της Ευρωπαϊκής Ομάδας του Ευρωπαϊκού Τίμ της Ευρωπαϊκής Αποστολής, καθώς και, της, και αξιολόγηση της επιχείρησης Μινουσμά. Δυστυχώς έγινε εκ του μακρόφεν, γιατί δεν μπορέσαμε να συναντήσουμε τους διοικητές της αποστολής Μπαρκάν. Όμως μπορέσαμε να κάνουμε μια αξιολόγηση και της αποστολής αυτής παρόλα αυτά και η συνολική εικόνα είναι θετική παρά τις ε, εξαιρετικές δυσκολίες. Topic that uh, Θα μπορέσουμε να μιλήσουμε για ένα πολύ σημαντικό θέμα, το θέμα της περιφερειοποίησης των αμυντικών, συγγνώμη, των προσπαθειών για την εξασφάλιση της ε, ασφάλειας ε, στο Σαχέλ. Ασχοληθήκαμε και κατά τη διάρκεια της αποστολής μας στο Μαλί με το θέμα αυτό. Συζητήσαμε επίσης διαμακρών με τις ε, συμμαχικές ειρηνευτικές δυνάμεις και με τα διάφορα μέρη που συμμετέχουν στην ειρηνευτική προσπάθεια ε, υπό την αιγίδα του πρέσβη της Αλγερίας, στο Μαλί δηλαδή διότι σε αυτή τη σύνθεση συναντώνται και μπορέσαμε επίσης να συναντήσουμε Ευρωπαίους διπλωμάτες των διαφόρων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που είναι διαπισταυμένοι στο Μαρίο. Επίσης λάβατε μια γραπτή έκθεση από τον κύριο Χαβιερνάτ που έμεινε λίγο περισσότερο στο Μαλί και ταξίδεψα και σε περισσότερα σημεία. Πήγε και στην Ήπεθρο. Δυστυχώς σήμερα δεν θα είναι μαζί μας. Γι' αυτό ζήτησε να παραταθεί γραπτή διαδικασία και η γραπτή διαβούλευση. για την έκθεσή μας επί της αποστολής στο Μαλί. Νομίζω σωστό θα ήταν να παραταθεί αυτό το διάστημα. Θέλω να δώσω το λόγο στον κύριο Νάρτ στις αρχές της επόμενης συνεδρίασής μας τον Οκτώβριο για να μας μιλήσει για τα πορίσματά του. Το πρόβλημα είναι όμως ότι πρέπει να βασιστούμε σε κοινέ αξιολογήσεις που έγιναν και από την αποστολή της ΣΕΝΤΕ και από την αποστολή της ΑΦΕΤ. Βασικά ήταν κοινή αποστολή της ΣΕΝΤΕ και της ΑΦΕΤ μαζί. Και στις συζητήσεις που κάναμε κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στο Μαλή προσπαθήσαμε να προβληματιστούμε από κοινού, θα πρέπει να βασιστούμε στα πόρισμα του κυρίου Νάρτ και θα πρέπει να φτάσουμε σε συνένεση βεβαίως. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στους συμμετέχοντες. Ο κύριος Ντέιβιτ Μακάλιστερ ήταν ένας από τους σημαντικούς συμμετέχοντες ε, που εκπροσώπησε την Επιτροπή ΑΦΕΤ. Έχετε το λόγο. Ε, Κυρία Πρόεδρε, δεν ζήτησα να πω κάτι, αλλά συμφωνώ απόλυτα με αυτό που λέτε. Αυτό αυτή, αυτή την επιτροπή. Πιστεύω ότι ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη και πιστεύω πως παρότι κάποιες συναντήσεις ακυρώθηκαν λόγω προβλημάτων στα σύνορα μεταξύ Μάλι και με Βρυτανίας, είχαμε ενδιαφέρουσα συζήτηση στην πρωτεύουσα Μπαμάκο. Με εντυπωσίασε το πως η εκπαιδευτική αποστολή προχωρά με τους Αφρικανούς στρατιώτες όχι μόνο από το Μάλι αλλά και από τις γειτονικέ χώρες ήταν μια πολύ αποδοτική επίσκεψη πιστεύω και έστειλα τα σχόλια μου επί της έκθεσης ήδη στη γραμματεία και πιστεύω πως πρέπει να κάνουμε μια συζήτηση εις βάθος όποτε αυτό είναι δυνατόν θα με ενδιαφέρει επίσης να ακούσω ε, αυτά που έχει να πει ο κύριος Νάρ. Ναι, ασφαλώς, συμφωνώ μαζί σας θα ήθελα να προσθέσω κάτι. Συνήθως δεν εξυμνώ τόσο εύκολα τα πράγματα, αλλά εντυπωσιάστηκα από το γερμανικό προχείρο νοσοκομείο εκεί. Υπάρχει ένα συμμετέχον ακόμα στην αποστολή, η κυρία Ντρογεύσκη ήθελα να πω αυτό που είπε και η, προε... η Προεδρεύουσα μόλις. Η επίσκεψη στο νοσοκομείο, το οποίο διευθύνεται από Γερμανούς στρατιώτες, πιστεύω πως αυτό που είδα εκεί ήταν ένας απίστευτος επαγγελματισμός στην εφοδιαστική όσο και στην εφαρμογή. Με αποτέλεσμα οι Γερμανοί στρατιώτες να, να έχουν δημιουργήσει με επιτυχία ένα τόσο μεγάλο ιατρικό κέντρο. Και πιστεύω επίσης ότι η επίσκεψη ήταν πολύ καλά προετοιμασμένη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ την... Θα ήθελα να ευχαριστήσω και τις δύο γραμματείες για την προετοιμασία της επίσκεψης αυτής. σημειώθηκε μια μεγάλη επίθεση και όλες οι κρατικές αρχές εστίαζαν στην επίλυση του προβλήματος της περίθαλψης των θυμάτων. Ωστόσο όλα έγιναν με ασφάλεια και πολύ επαγγελματικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ ασφαλώς θα ήθελα να συνεχίσω τη συζήτηση. Το Σαχέλ είναι μια, ένα πολύ περίπλοκο θέμα και πιστεύω πως το Μάλι θα απασχολήσει τις συζητήσεις της ΣΕΔΕ τους επόμενους μήνες και στο απότερο μέλλον. Προσωπικά με ενδιαφέρει πολύ η προφορική έκθεση του κυρίου Νάρτ για την επίσκεψή του κατά τη συνέχεια της συζήτησης. Συγγνώμη. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για αυτό το μέρος η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η επόμενη συνεδρίαση οπότε ελπίζω να μπορέσουμε να συμφωνήσουμε για μια κοινή στάση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το επόμενο σημείο είναι η περιφερειοποίηση για τις αποστολές στα πλαίσια της ΚΠΑ στο Σαχέλ. Με μεγάλη μου χαρά θα ήθελα να παρουσιάσω τον κύριο Ζακ Φραντέλ, ο οποίος είναι διευθύνων του τομέα ολοκληρωμένου στρατηγικού σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης θα γίνει μια συνέχεια της προηγούμενης συζήτησής μας. Θα ήθελα επίσης να επενθυμίσω πως ήδη συναντήσαμε τον κύριο πρέσβη Ανχέλ Σάντα πριν από το θερινό διάλειμμα, ο οποίος παρουσίασε ήδη κάποιες απόψεις και προοπτικές της περιφερειοποίησης των εγχειρημάτων ασφάλειάς μας και τώρα ήρθε η ώρα για τον κύριο Φράνταν να παρουσιάσει τις απόψεις του. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ για αυτή την ε, πρόσκληση που μου κάνετε για να μιλήσω για το θέμα της ε, περιφερειοποίησης. Θα γίνει και άλλη παρουσίαση για το Μαλή. Το Μαλί είναι στο, στην καρδιά αυτή της περιφερειοποίησης. Ε, θα σας εξηγήσω σχηματικά αυτή την ε, έννοια. Ε, το γενικό τροπλαίσιο της περιφερειοποίησης. δεύτερον, η πιθανή στόχη αυτής της περιφερειοποίησης. Και τέλος, περιγραφή Πώς θα μπορούσε να γίνει αυτή η περιφερειοποίηση το γενικό πλαίσιο να υπενθυμίσω ότι η σταθερότητα στη Σαχέλ είναι στρατηγική σημασία για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα κράτη-μέλη. Ε, de facto, μια μεγαλύτερη σταθερότητα στι χώρε αυτέ ε, τη περιοχή θα συνεισφέρει στην ευρωπαϊκή ασφάλεια και θα επιτρέψει να υπάρξει θετική επίπτωση ε, στου κινδύνου που αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά αυτό χρειάζεται μια συνεχή δράση και μια δέσμευση απαρασάλευτη μεταξύ ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των πέντε χωρών του Σαχέλ. Τσάντ, Μαφριτανία, Μπουρκίνα Φάσο, Νίγηρας και Μαλή. Υπάρχει ε, το πέντε Σαχέλ. Είναι μια νέα δομή η οποία δημιουργήθηκε. Θα πρέπει αυτή η εταιρική σχέση να εντατικοποιηθεί με τα κράτη-μέλη και με του υπόλοιπου διεθνεί οργανισμού που είναι παρόντε, καθώ και με την ε, διαδικασία που είναι ήδη εν εξελίξη. Στο θέμα της, ε, που μας ενδιαφέρει, την ασφάλεια και την άμυνα, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αυξήσει τις, ε, το εθνικό δυναμικό του Σαχέλ, αλλά και τη συνεργασία ε, ανάμεσα σε αμυντικές δυνάμεις ούτω ώστε να βελτιώσουμε το δυναμικό απέναντι στι απειλέ και στου κινδύνου που αντιμετωπίζουν οι χώρε αυτέ. Όπω ε, υπόθηκε, θα πρέπει να δώσουμε και τον απαραίτητο χώρο σε περιφερειακέ πρωτοβουλίε, κυρίω ε, του G5 Σαχέλ, που θα είναι στον πυρήνα της προσπάθειας ε, περιφερειοποίησης. Αυτό επαναδιατρανώθηκε το, από του Υπουργού Άμυνα τον Ιούνιο όπου ε, ζητήθηκε από την Υπηρεσία Εξωτερική Δράση να παρουσιαστεί ένα σχέδιο που θα επιτρέψει στα κράτη-μέλη να δεσμευτούν απέναντι στο Σαχέλ ε, μέσω και των ε, αποστολών περιφερειοποίηση. Αυτή η έννοια αναπτύχθηκε και θέλω να σας παρουσιάσω το πλαίσιο μέσα στο CSDP θα ενταχθεί. Η σχέση ανάμεσα στην εξωτερική και εσωτερική ασφάλεια και σε τομείς όπως το οργανωμένο έγκλημα ε, το λαθρεμπόριο, η τρομοκρατία. Είναι ένα σημαντικό πλαίσιο για πιθανές ε, επιχειρήσεις της ΚΠΑ. Η δέσμευσή μας απέναντι στα ΧΕΛ θα πρέπει να συνδεθεί με τις προσπάθειές μας στη Λιβύη, ε, στο της Αφρικής και στην Δυτική Αφρική. Η περιφερειοποίηση των αποστολών ε, ΕΠΑ θα επιτρέψει ε, να βελτιώσουμε την ασφάλεια και να αυξήσουμε τις αμυντικές δυνατότητες των χωρών Σαχέλ, δίνοντας σημαντική συνεισφορά ε, και αυτές οι χώρες με την πλευρά τους για την ασφάλεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν τρεις αποστολές ΕΠΑ στη Σαχέλ, δύο πολιτικές, στο Μαλί και στον Νίγηρα και μία ε, στο Μαλί στρατιωτική. Δηλαδή τρεις αποστολές στο Σαχέλ. Ο, ο στόχος της περιφερειοποίησης είναι να αξιολογήσουμε τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα ομαδοποιήσουμε τις προσπάθειές μας ε, για τις χώρες αυτές του G5, ειδικά εκεί που δεν έχουμε αποστολές ΕΠΑ, δηλαδή Μπουρκίνα Φάσο, Τσάντ και Μαυριτανία. Η ανάπτυξη των επιπλέον προσπαθειών στις τρεις αυτές χώρες ε, θα γίνουν, ε, και αυτό το τονίζουν τα κράτη-μέλη, ε, με βάση, ανάλογα με την εντολή που θα έχει η κάθε επιχείρηση. Αυτό το λαμβάνουμε υπόψη μας για να γίνει αυτή η περιφερειοποίηση. Ε, δεν θα πρέπει να αποδυναμώσουμε αυτό που ήδη γίνεται και δίνει αποτελέσματα. Αυτό σημαίνει καλό συντονισμό με τα κράτη-μέλη που είναι παρόντα στι ε, χώρε τη περιοχή, την Κομισιόν, τον ειδικό εκπρόσωπο τη Ευρωπαϊκή Ένωση για το Σαχέλ, του διεθνεί εταίρου και φυσικά και τι χώρε τη ε, περιοχή αυτή. Τρίτο και τελευταίο σημείο, οι στόχοι και οι προσπάθειες των, της περιφερειοποίησης ε, των επιχειρήσεων ΕΠΑ είναι προωθούν τρεις στρατηγικούς όρου. Να βελτιώσουμε τις ε, εθνικές προσπάθειες και δυναμικό των χωρών, να βελτιώσουμε την ε, διασυνορική συνεργασία ε, περιφερειακές και τις περιφερειακές δομές περιφερειοποίησης, ειδικά των χωρών G5 Σαχέλ. την περασμένη Πέμπτη στο ΚΟΠ συζητήσαμε την έννοια της περιφερειοποίησης και θα ξανασυζητηθεί τον Οκτώβριο αφού υποβληθεί στην συναφή ομάδα, στις συναφές, ομάδες ε, και που θα γνωμοδοτήσουν και αυτή τη στιγμή τα κράτη-μέλη επίσης πούν την άποψή τους. Γενικά ε, θα έχουμε τρεις φάσεις στην περιφερειοποίηση αυτή. Στην πρώτη φάση θα δημιουργήσουμε ένα δίκτυο εμπειρογνωμόνων που για το Μαλή θα έχει ένα κέντρο ε, περιφερειακής διοίκησης και σε κάθε μία από τις χώρες αυτής ε, θα στις δικές μας χώρες θα έχουμε μάλλον έναν αξιωματικό συνδέσμο που είναι υπεύθυνοι ε, για θέματα άμυνας ή ασφάλειας που θα μας επιτρέψουν να κάνουμε αξιολόγηση των αναγκών και του δυναμικού που θα πρέπει να ανοιχθεί, ε, τι βοήθεια μπορούμε να δώσουμε στις χώρες, καθώς και να αναπτύξουμε ένα περιφερειακό σχέδιο επιχειρησιακής φύσεως τύπου ΕΠΑ για τις χώρες αυτές που θα επιτρέψει αυτή τη στιγμή αναπτυχθεί και υπάρξουν και τα απαραίτητα εργαλεία, να γίνει μια καλή, ε, ένας καλός συντονισμός της ε, συνολικής ε, δραστηριότητας Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την πρώτη φάση, τη δημιουργία δηλαδή του δικτύου εμπειρογνωμόνων, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι με, αυτό το, αυτό το δίκτυο μέχρι τον Ιούνιο του 2017. Δεύτερη φάση επιχειρησιακή φάση. Άμεσε δράσει τη ΕΠΑ, δηλαδή εκγύμναση που θα μπορούσε να γίνει για να δούμε τι δυνατότητε έχουμε, ε, ε, και να βοηθήσουμε τι πέντε χώρες ε, του G5. Ε, θα βοηθήσουν τα άτομα τα οποία είναι επιτόπου με βάση ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα ανάλογα με τη δυνατότητα απορρόφησης με βάση τα όσα εντοπίσαμε στη φάση της αξιολόγησης που κάναμε. Αυτό που υπόθηκε προηγουμένως είναι σωστό. Δηλαδή, τον Ιούλιο διαπιστώσατε κάποια πράγματα με αυτά που σας λέω. Δηλαδή, κάναμε ένα τεστ ε, περιφερειοποίησης για να δούμε ε, πώς μπορούμε να εντοπίσουμε καλύτερα, να γυμνάσουμε τους ανθρώπους και να βασιστούμε στα όσα έχουμε. Η τρίτη φάση θα έρθει αργότερα και με βάση τα όσα θα έχουμε καταφέρει θα δούμε εάν θα πρέπει να επεκτείνουμε την παρουσία ΕΠΑ στις χώρες ε, Σαχέλ. Φυσικά όλα αυτά εξαρτώνται από την ε, πρόθεση των κρατών μελών. Και ανάμεσα στην ε, πρώτη φάση και τη δεύτερη φάση, δηλαδή αφού κάνουμε την αξιολόγηση, τα κράτη-μέλη θα αποφανθούν εάν χρειαστεί να περάσουμε στη δεύτερη φάση ή αν θα πρέπει να αναθεωρήσουμε το συνόλο του μηχανισμού αυτού. Δηλαδή έχουμε μία βαθμιά προσέγγιση υπέρ των χωρών αυτών του G5. Κλείνω εδώ λέγοντας ότι προς το παρόν τίποτα δεν έχει αποφασιστεί γιατί θα πρέπει τον Οκτώβριο να ε, αποφανθούν τα κράτη-μέλη. Παραμένω σε διάθεσή σας για οποιαδήποτε ερώτηση μου υποβάλλατε. Oh. Σας ευχαριστούμε. Παρακαλώ, αν θέλετε, πάρετε το λόγο. Στο μεταξύ, να κάνω κι εγώ μια ερώτηση. Είναι πολύ παίκτε στην περιοχή του κόσμου. Πιστεύετε ότι όλοι προτίθεται να λάβουν υπόψη αυτή την περιφερειακή προσέγγιση για την ασφάλεια Πρόκειται για μια πρωτοβουλία μόνο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα εφαρμοστεί στα πλαίσια των διμερούς τη Ένωση ε, με τρίτες χώρες ε, σε αυτή την περιοχή. Α, ο Χαριστούμε, Ευχαριστούμε, Πρόεδρε. Ε, νομίζω ότι για αυτή την έννοια της περιφερειοποίησης υπάρχει σχετική ομοθυμία. Είναι λογικό και ε, σίγουρα θα συνεπάγεται και εξορθολογισμό των ε, κατακαιρματισμένων αυτή τη στιγμή προσπαθειών στην περιοχή της Αχέλ. Για να ε, επισέλθω και σε λεπτομέρειες, πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση σε σχέση με τον τρόπο εκτέλεση του σχεδίου μας, κυρίως για τη δεύτερη φάση που προαναφέρατε, επιχειρήσεις ε, κατάρτισης εκπαίδευσης σε σχέση με υφιστάμενες επιχειρήσεις ε, ΕΠΑ. Ξέρετε ότι οι εθνικές και ενδοεθνικές ευαισθησίες είναι, έχουν πολύ έντονη παρουσία. Δεν ξέρω αυτά που γίνονται τώρα στο Μάλι, στην Ιγυρία, αν ε, τελικά είναι κατάλληλα για να αναπτυχθούν επιχειρήσεις εκπαίδευση στα πλαίσια του G5. Θα πρέπει να γνωρίζουμε τις προθέσεις των ΜΕΝ και των ΔΕ. Όσες χώρες του G5 δεν έχουν επιτόπου επιχειρήσεις, φαντάζομαι θα θέλουν να έχουν στην επικράτειά τους συγκεκριμένε επιχειρήσεις εκπαίδευσης του δικού τους προσωπικού που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του προσωπικού τους. Ε, γι' αυτό δεν είμαι και σίγουρος ότι μια συγκεντρωτική επιχείρηση ε, στο Μάλι θα οδηγήσει σε ενσωμάτωση όλων σε έναν μηχανισμό. Δεν το δηλώνω αυτό, απλώς ε, αναρωτιέμαι πώς θα εξελιχθεί αυτή η ιδέα. Ε, σε αυτές τις απαρχές της περιφερειοποίησης, αυτή την ευρωπαϊκή προσπάθεια θα πρέπει να έχουμε feedback από το G5, δηλαδή να ξέρουμε ποιος είναι ο απόϊχος ε, αυτών των προτάσεών μας. Μην ξεχνάτε ότι στις επιτόπιες δυναμίες υπάρχει ανομοιομορφία. Έχω στο κατά νου συγκεκριμένα το μάλι. Ε, πρόκειται για ένα στρατό υπό διάλυση θα έλεγα, ανοργάνωτο, ε, που μετά την τζιχαντιστική επίθεση του 2012 και των αρχών του 2013 ε, είχε κλονιστεί. Ε, Είδητε τη Μαυριτανία. Πολλές από τις δυνάμεις ασφαλείας αναδιαρθρώθηκαν και καταβάλλονται σημαντικότατες προσπάθειες και οι ανάγκες δεν είναι απαραίτητα της ίδιας φύσης σε σχέση με αυτά που επιδιωκούν στο Μάλι. Ξαναλέω, είναι ανομοιόμορφες οι περιστάσεις Καλά, καλή ιδέα ακούγεται αυτή της περιφερειοποίησης, επί της αρχής να την υποστηρίξω. Φαίνεται λογική ιδέα, όμως προσοχή, είναι ε, πολύ διαφορετικές οι καταστάσεις που επικρατούν στις χώρες και άρα ε, προϋποθέτουν και διαφορετικές ε, απαντήσεις. Προσοχή λοιπόν. Καταλαβαίνω, λέει η Πρόεδρος, ε, από ό,τι βλέπω ότι κανείς δεν θέλει το λόγο προς το παρόν. Οπότε, παρακαλώ, ε, ε, σχολιάστε τις ε, παρεμβάσεις των βουλευτών και ίσως κάνουμε δεύτερο γύρο. Ο εισηγητής, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Ε, σχετίζονται με τον πυρήνα των προτάσεων μας σε σχέση με τις πιθανές ατέλειες και τις δυναμικότητε που υπάρχουν επί ναι, ναι, θα πρέπει όλα αυτά να τα εξετάσουμε προσεκτικά. Και μιλήσατε για ε, αναχώρα προσέγγιση, δική προσέγγιση. Βεβαίω, ε, χαίρονται ναι, ε, στο Τσάτ, στη Μαυρετανία και στη Μπούρκινα Φασό να έχουν εμπειροχνόμενε από τα κράτη-μέλη. Αλλά καλό θα είναι να ενοποιηθεί η δράση μα σε πολλού τομεί. Δεν μιλάω μόνο για ΕΠΑ. Ε, υπάρχουν και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι συνομιλητές μας αυτές οι ένοπλες δυνάμεις μας επιτρέπουν να υλοποιήσουμε το σχέδιό μας λαμβάνοντας υπόψη αυτά που μας είπε ο κύριος Ντανζάν, δηλαδή λαμβάνοντας υπόψη και τα εθνικά συμφέροντα σε σχέση με τις απειλές. Υπάρχει υποστήριξη λοιπόν και αυτό το είδαμε και στη Σύνοδο ανάμεσα στην είπα εκπρόσωπο ε, και το ε, χώρες του G5 τον Ιούνιο, γιατί ετέθη αυτό το ζήτημα και υπήρξε πλήρης υποστήριξη για αυτή την έννοια. Φυσικά με εφαρμοστικά μέτρα που θα προσδιορίσουμε εκ των υστέρων ε, ως τους λεπτομέρειες. Τώρα, για τις διεθνείς οργανώσεις, κυρίως όταν μιλάμε για το Μάλι, αλλά και για την Ιγυρία και για άλλους εταίρους μας, και για το τσάτ το ίδιο ε, ισχύει. Συμφωνούν με αυτά που προτείνουμε για την πρώτη φάση. Ε, μπορεί να υπάρξει μια νεολογική προσέγγιση, παρόλα αυτά κανείς δεν μπορεί να προβλέψει πριν να γίνει συνολική αξιολόγηση πώς ακριβώς θα προβούμε στο στάδιο 2. Οπότε για να δώσω συγκεκριμένη απάντηση, ναι, προσυπογράφουν όλοι ε, το στόχο αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δούμε αυτή η δέσμευση τι έμπρακτα αποτελέσματα θα έχει, είναι υψηλέ οι προσδοκίε ε, ασφαλώ και θα δούμε ε, σε ποιε μπορούμε να ανταποκριθούμε και ε, πού μπορούμε να αντισταθμίσουμε τυχόν ελλείψεις. Στα πλαίσια του G5 έχουμε πέντε κράτη με κοινά συμφέροντα αλλά και διαφορετικές, διαφορετικούς στόχους. Γι' αυτό και μίλησα για ε, διασυνοριακή συνεργασία, γιατί δεν είναι, οι ανησυχίε ε, διαφέρουν από χώρα σε χώρα, τα, ε, τα συμφέροντα διαφέρουν από χώρα σε χώρα, φυσικά. Για την περιφερειοποίηση, τον Οκτώβρη περιμένουμε τοποθέτηση των κρατών μελών. Υπάρχει ένα κενό και προσπαθούμε να τα αποκλειστούμε σε αυτό. Υπάρχει στρατηγική του, τη, στην περιοχή του Σαχέλ και με την ε, στρατηγική περιφερειοποίηση ε, θα μπορούσαμε να αξιοποιήσουμε τους ε, αξιωματικούς συνδέσμους, είτε πρόκειται για ΕΠΑ, είτε μιλάμε για άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα δούμε πού έχουμε τα μέσα για να ε, έχουμε ε, μέσω παραδείγματος χάρη καταπιστευμάτων ή έκτακτων χρηματοδοτικών μέσων πώς μπορούμε να ενισχύσουμε τις προσπάθειε μας και τις επιχειρήσεις ε, στο πλαίσιο της ΕΠΑ. Βλέπετε αυτή είναι η προσθέμενη αξία ε, της περιφερειοποίησης. Φυσικά το περιεχόμενο της δεύτερη φάσης θα το προσδιορίσουμε στη συνέχεια όπω σα έλεγαν τα κράτη-μέλη. σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να γίνει πρώτη εξολόγηση και μόνο να διαπιστωθεί η ανάγκη θα οδηγηθούμε σε αυτό το δεύτερο στάδιο και όπως είπαμε ε, σε τοπικό επίπεδο και σε σχέση με συγκεκριμένες απειλές σε εθνικό επίπεδο θα αναπτύξουμε λύσεις και έτσι το σχέδιο περιφερειοποίησης θα περάσει σε επιχειρηματικό στάδιο, επιχειρησιακό στάδιο και θα βασιστούμε φυσικά στον κορμό της ΕΠΑ. Δεν θέλουμε να καταστήσουμε τις επιχειρήσεις, θέλουμε να αξιοποιήσουμε τις εμπειρίες μας, ε, ούτως ώστε να μην έχουμε τάγματα ε, στρατιωτών ή αστυνομικών. Όχι, στοχευμένες δράσεις ε, επιδιώκουμε για να βοηθήσουμε αυτά τα κράτη, ούτως ώστε να μεγιστοποιήσουμε το δυναμικό που έχουμε ήδη αναπτύξει ανάλογα με την ικανότητα απορρόφησης των κρατών μελών. Να δούμε σε ποια προς μία κατεύθυνση θέλουν να αναπτυχθούν. Ε, ε, ε, ιεραρχούν με τον ίδιο τρόπο τις προτεραιότητες τους σε σχέση με την πρώτη φάση. Σε σχέση με το Μάλι, ε, αυτά έχουμε κάνει μέχρι σήμερα και γι' αυτό το προτείνουμε. Έχουμε τον παράγοντα χρόνο και το παράγοντα εξοικονόμηση και αποτελεσματικότητα. Για το χρόνο, γιατί έχουμε δύο ε, επί επιτόπου. Εάν θέλουμε συντονισμό χωρίς να επανεφεύρουμε το, το, το, τροχό θα πρέπει να συντονίσουμε τη δράμη σας και μετά. Έχουμε λοιπόν ε, ε χάρη στο συντονισμό ε, αυτών των δύο στρατιωτικών ε, της στρατιωτικής και μη στρατιωτικής επιχείρησης σε μέγιστη αξιοποίηση των δυνατοτήτων μας πως ε, τώρα θα αντιποκριθούμε στους συγκεκριμένου ε, στόχους και τα συμφέροντα των ε, χωρών της ομάδας G5 όταν γίνει ε, ε, χαρτογράφηση των επιχειρησιακών αναγκών θα δούμε στην Μπούρκινα Φάσο και στο Μάλι δεν έχουμε τις ίδιες ε, το, ούτε και στη Μαυρετανία υπάρχουν ιδιαιτερότητες και Φυσικά θα υπάρξει συνεργασία των πέντε χρονών, αλλά θα λάβουμε δεόντως υπόψη την περιφερειακή, την τοπική διάσταση. Για να αντιμετωπίσουν αυτές οι χώρες ε, τις απειλές ε, ε, ίσως μην χρησιμοποιήσουμε την ε, ΕΠΑ, να χρησιμοποιήσουμε άλλα ε, όργανα. Σε κάθε περίπτωση θα χρειαστεί συντονισμό ε, και κάποια κράτη ίσως διαπιστώσουν ότι χρειάζονται εκπαίδευση επιτόπου. Μιλήσατε για τις κοινωνικές ευαισθησίες. Κυριολεκτικά το καταλαβαίνω ότι υπάρχουν αυτές οι ευαισθησίες. Οι απειλές είναι ε, κοινέ αλλά και διαφορετικές. Οπότε, στην πρώτη φάση αυτό θα κάνουμε. Θα κάνουμε την ανάλυση ούτω ώστε ε, να καταθέσουμε συγκεκριμένες προτάσεις στα κράτη-μέλη. Μόλις καταλάβουμε, μόλις αναλύσουμε τι χρειάζεται ε, σε κάθε χώρα για να αντιμετωπίσουμε ε, τους κινδύνους και ο βεβαίως να θωρακίσουμε τα σφαίρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης κύριε Ευχαριστώ για τις εξηγήσεις σας. Θέλω να επανέλθω στην πρώτη φάση της περιφερειοποίησης για την ομάδα για το δίκτυο αυτό εμπειρογνωμόνων. Είχαμε εκφράσει μια σχετική ανησυχία στην Υποεπιτροπή και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων εδώ και αρκετό καιρό. Ότι θα πρέπει οι αντιπροσωπείε δηλαδή τη Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουν του δικού εμπειρογνώμονε για θέματα ασφάλεια και άμυνα ειδικά στις αντιπροσωπείες των χωρών όπου υπάρχουν αποστολές ΕΠΑ, αλλά και σε αντιπροσωπείες που βρίσκονται σε ζώνες κρίσης και που έχουν προτεραιότητα για λόγους ασφάλειας. Υπάρχει περίπτωση αυτή, αυτό το δίκτυο εμπειρογνωμόνων να αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο, δηλαδή πιο μόνιμο, ή είμαστε ε, στα πλαίσια μιας ad hoc αποστολής, ε, πολύ εξειδικευμένης, που δεν θα βασιστεί στις ε, ε, που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε διάφορες χώρες, αλλά θα βασιστεί κυρίως στις δομές που υπάρχουν στο Μπαμάκο. Θέλετε να σχολιάσετε. Θέλω να θέσω κι εγώ μία επιπλέον ερώτηση. όπως είπα και πιο πριν, κατά τη διάρκεια της παραμονής μας στο Μάλι, έλαβε χώρα μία επίθεση σε ένα στρατιωτικό σύνδεσμο κοντά στα μαυριτανικά σύνορα. Οι επιθέμενες μονάδες ήταν καλώς εξοπλισμένες, ήρθαν με οπλισμένα οχήματα, πολύ πιθανόν από την επικράτεια της Μαυριτανίας και από ό,τι φαίνεται μπόρεσαν να αντιμετωπίσουν επιτυχώς τα στρατεύματα του Μάλι. Τι χρειάζεται μετά από μια τόσο μακρά δραστηριοποίηση. Ποια είναι η κατάσταση των στρατών των πέντε αυτών περιφερειακών χωρών. τι σενάριο θα πρέπει να υλοποιήσουμε για να ενδυναμώσουμε τους στρατούς αυτούς πραγματικά και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να καταπολεμήσουν επιτυχώς την τρομοκρατία. Καταρχά, να απαντήσω στο ερώτημα του κ. Ντανζόν, που είναι και πιο απλό για μένα. Να απαντήσω στο ερώτημα του κ. Ντανζόν. Ε, θα μπορούσα να είχαμε μιλήσω λίγο περισσότερο για την αρχή αυτή των αξιωματικών συνδέσμου που είναι είτε στρατιωτικοί ή μη στρατιωτικοί και που θα εντάσσονται στις αντιπροσωπείες και που θα έχουν το ρόλο που μόλις περιγράψατε. Ε, κάνουμε την ίδια διαπίστωση ε, ότι πρέπει ε, ειδικά σε περιοχές ε, κρίσης να έχουμε αυτή τη δυνατότητα ε, και δημιουργούμε αυτό το δίκτυο γιατί υπάρχει αυτή η έλλειψη. Αυτό το δίκτυο λοιπόν αξιωματικών συνδέσμου θα παραμείνει σε όλη τη φάση της ε, προσπάθειας περιφερειοποίησης, σε όλη τη φάση δηλαδή που θα αναπτύσσονται οι επιχειρήσεις ΕΠΑ. Αν προκύψει κάτι άλλο μετά σε μια μεταγενέστερη φάση, τότε θα θέσουμε το ερώτημα. Αλλά τώρα θέλουμε να δράσουμε γρήγορα με τα μέσα που έχουμε. Αυτό λοιπόν έχουμε προβλέψει. Ε, τώρα, τι πρέπει να κάνουμε, κυρία Πρόεδρε, είναι περίπλοκο αυτό το ερώτημα. Δεν είμαι εμπειρογνώμονα και δεν μπορώ να απαντήσω συνολικά στο ερώτημα. Θα παραμείνω στο δικό μου το τομέα που ξέρω, δηλαδή την ΕΠΑ ε, την αποστολή, ας πούμε, ε, στο Μαλί και το ρόλο που έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω των, του ειδικού εκπροσώπου και της αντιπροσωπείας μας. Γιατί ε, υπάρχουν πολλαπλά προβλήματα για την κυβέρνηση του Μαλί. Έχουμε το πρόγραμμα ΠΑΡΣΕΚ, πρόγραμμα βοήθειας ε, μέσω ε, των κονδυλίων του καταπιστεύματος αυτού, που δεν είναι μια δράση μόνο στρατιωτική, είναι μια δράση σε πολλά μέτωπα ό,τι κάνουμε προσπαθούμε να το κάνουμε στον τον καλύτερα. Μην ξεχνάτε όμως ότι από πλευρά μας, ε, όπως είπε ο κ. Ντονζό, έχουμε να κάνουμε με ένα στρατό ο οποίος είναι υποδιάλυση, ο οποίος προσπαθεί να ξαναδημιουργηθεί απέναντι σε μια απειλή η οποία αλλάζει μορφή συνέχεια. Ε, θα πρέπει να μιλήσουμε και με άλλους ανθρώπους που είναι πιο παρόντες στο στατιωτικό μέτωπο. Ε, εγώ αυτά που μπορώ να σας πω είναι ότι δεν θα πρέπει να μειώσουμε τη δράση μας στον τομέα των επιχειρήσεων ΕΠΑ, γιατί δίνουν αυτές οι επιχειρήσεις καρπούς. Όταν βλέπετε, βλέπουμε τέτοιες επιθέσεις όπως αυτή που αναφέρατε, ε, είναι σημαντικό να έχουμε αυτές τις, αυτό το δυναμικό, αυτές τις δράσεις. Ε, και ο, θα πρέπει ο στρατός του Μαλή να έχει τη δυνατότητες να αντιμετωπίσει τέτοιες προκλήσεις. Ο κ. Παπαδάκης. Ε, thank um, President. Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε θα ήθελα να πω πως αναφερόμαστε σε μια πολύ επικίνδυνη εξέλιξη. Μιλούμε για μια επέμβαση σε περιφερειακό επίπεδο, το οποίο σημαίνει μια κλιμάκωση των υπεριαλιστικών παρεμβάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αφρική. Η κατάσταση είναι ρευστή, πολύ ρευστή σε όλη την περιοχή και φυσικά θα έπρεπε να έχετε κατά νου πως φέρεται μεγάλη ευθύνη. για αυτή την κατάσταση. Επειδή δεν μπορούμε να πιστέψουμε την δικαιολογία που αναφέρεται για τη δημιουργία, για την παροχή εκπαίδευσης του στρατούς, ο κύριος λόγος της παρέμβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η ανάπτυξη των σχεδίων των μεγάλων μονοπωλίων εκεί σε έντονη σύγκρουση με τις Ηνωμένε Πολιτείε και την Κίνα επειδή αυτοί είναι οι δύο σημαντικοί παράγοντες στην περιοχή και τα ευρωπαϊκά μονοπόλια θέλουν να παρέμβουν επίσης για να ελέγξουν ένα μέρος των πλούσιων πόρων των πέντε χώρων αυτών. Έχετε λοιπόν κατά νου την όλη κατάσταση, την όλη ιστορία του Μάλι, της Λιβύης και όλες τις επεμβάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα ήθελα να ξέρω ποια θα ήταν οι πρώτες αντιδράσεις των ΗΠΑ και της Κίνας μετά από την δήλωση αυτή Τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ε, ευχαριστώ, ο κύριος Φραντόν. Ευχαριστώ για το ερώτημά σα. Ήρθαμε σε επαφή με τους εταίρου. Ήρθαμε σε επαφή με τους Αμερικάνους εννοώ οι οποίοι είναι παρόντες, ε, πολύ παρόντες στις χώρες ε, του Σαχέλ και στο Μαλί και στο Νίγηρα και προωθούν δράσεις που μας ενδιαφέρουν και εμάς στον Ήγηρα, εκείνοι ασχολούνται με το στρατό μαζί με, τις, ε, με άλλες χώρες, ε, ενώ εμείς ε, σε επίπεδο ΕΠΑ είμαστε πολύ πιο περιορισμένοι. Κάνουμε κατάρτιση, παρέχουμε εκπαίδευση στο στρατό. Οι Αμερικανοί έχουν τη δική τους παγκόσμια στρατηγική, την ξέρετε. Ε, πάντως εμείς στο επίπεδο της ΕΠΑ ε, λειτουργούμε με διαφανή τρόπο. Θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα στι δυνάμει τη χώρα των χωρών αυτών να παίξουν, τις στρατιωτικέ δυνάμεις δηλαδή, να εξασφαλίσουν την εδαφική ακαιρεότητα τη χώρα. Ε, για την ε, συνεργασία με, την, ε, με τη ΣΥΠΑ στα πλαίσια τη ΕΠΑ πρέπει να σα ομολογήσω η συνεργασία αυτή λειτουργεί καλά. Σε ό,τι αφορά την Κίνα, οι δράσει του στα πλαίσια τη ενίσχυση του στρατιωτικού ή μη δυναμικού είναι αρκετά δύναμη στη χώρα αυτή. Για μα δεν είναι καν συνομιλητή η Κίνα στους τομείς τουλάχιστον που δραστηριοποιούμαστε. Στους άλλους τομείς που εσείς αναφέρατε, δεν είμαι ο καταλληλότερος άνθρωπος για να σας απαντήσω. Ζητώ συγγνώμη γι' αυτό. Αλλά ούτως ή άλλως, κάναμε τις απαραίτητες διπλωματικές προσπάθειες, ούτως ώστε η δική μας δράση στα πλαίσια της ΕΠΑ, να μην είναι εις βάρος των δεσμεύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά υπέρ μιας συνεργασίας και σε διεθνές επίπεδο για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα τα οποία έχουμε εντοπίσει, τα οποία έχουν διεθνή διάσταση. Είναι το μόνο που μπορώ να πω στην ερώτησή σας. Ευχαριστώ. Oh, Ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου άλλη μια ερώτηση να κάνω. Έχουμε αντιλήσει διδάγματα από την επιχείρηση Μπακόν. Στην περιοχή αυτή. κυρίως ε, στα πλαίσια των διοικητών των επιχειρήσεων. Διαπιστώσαμε ότι υπήρχαν διαφορές ως προς τις εντολές. Τι περαιτέρω μπορούμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις μας επιτόπου Από την αρχή της επιχείρησης και της στρατηγικής ε, του Μάλι για την περιοχή της Σάχελ είναι πολύ έντονη η παρουσία τρομοκρατικών οργανώσεων και είναι πολλά και πολυδιάστατα τα προβλήματα. Γι' αυτό σας ρωτώ, ποια δάγματα μπορείτε να αντιλήσετε από τις επιχειρήσεις μας μέχρι τούτο. Απάντηση από την ε, γαλλική παρουσία στη περιοχή της Αχέλ, μπορώ να σας πω ότι ε, είτε μιλάμε για τη μελλοντική περιφερειοποίηση, είτε μιλάμε για τις επιχειρήσεις ΕΠΑ, ε, είμαστε πολύ ικανοποιημένοι από την γαλλική παρουσία. Α, ναι, λέει πρόεδρος, ναι. Για την ίδια την επιχείρηση και την... το πώς εκτελήχθηκε, δεν είμαι αρμόδιος, ούτε ειδικό να σας πω ε, επικαλέσει το άρθρο 42.7 η Γαλλία, όπως είπατε. Και η Γερμανία ανέλαβε δέσμευση στο Μαλί. Αυτό θα λειτουργήσει ως παράδειγμα ίσως ε, και για άλλες οργανώσεις, ε, γιατί υπάρχουν κενά και σε επίπεδο παράδειγμα του χάρη. Μία ε, ενής λογική δράση, αν αποσιάσουν κάποιοι φορείς επιτόπου, ε, σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε σε παγρύπνηση και είναι ό,τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε εμείς στον τομέα της άμυνας, ε, γιατί πρώτα θα γίνει ανάλυση των αναγκών στην πρώτη φάση και μετά θα προσδιοριστεί η επιχείρηση στη δεύτερη φάση. Όταν αντιμετωπίζει εξωτερικές ή και εσωτερικές απειλές μια χώρα, ε, ε, δύσκολα μπορεί να καθησυχαστεί και πρέπει ε, να την καθησυχάσουμε και να την βοηθήσουμε να υπερπηδεί στις δυσκολίες. Και για να είναι βιώσιμη η επιχείρησή μας πρέπει να γίνει αυτή η ανάλυση των αναγκών. Ευχαριστούμε. Υπάρχουν άλλες παρατηρήσεις. Όχι. Μάλιστα. Ολοκληρώνεται και αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης. Σας ευχαριστούμε και ελπίζουμε να είστε παρόν σε μελλοντικές συνεδριάσεις της ΣΕΝΤΕ γιατί θα ανακύψει και πάλι το ζήτημα του Μαλή. Είναι όπως καταλαβαίνετε δύσκολο να γίνεται η έκθεση πεπραγμένων γιατί είναι περίπλοκη η κατάσταση και δύσκολα μπορούμε να καταλήξουμε σε συνένεση. Αλλά σίγουρα θα έχουμε καλά αποτελέσματα χάρη και στη συνεργασία μας. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, ε, παρακαλώ να ε, μείνετε στην αίθουσα. Έχουμε πάρα πολύ σημαντική συζήτηση που ακολουθεί. Στο μεταξύ, επιτρέψτε μου να σας πω πώς από τη συνεδρίαση που έγινε την 5η Σεπτεμβρίου θέλουμε να εγκρίνουμε τα πρακτικά κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης. Αν δεν γίνουν παρατηρήσεις, ε, προβληθούν ενστάσεις θα θεωρήσω ότι εγκρίνονται τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, Ζητώ συγγνώμη που δεν το ανέφερα. We wait just um, θα περιμένουμε για το δεύτερο πανελίστα λίγα λεπτά. Ladies um, Κυρίες και κύριοι, το επόμενο σημείο είναι η στρατιωτική άσκηση της Ρωσίας Κάφικας 2016 έγινε πρόσφατα και θα εξετάσουμε τις επιπτώσεις της ως προς την περιφερειακή ασφάλεια. Οι δύο διακεκριμένοι πανελίστες μας ε, είναι ο ενεργή επικεφαλής ε, της, του κλιμακίου της ε, Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, ο κύριος Γέχορ Μπόσοκ, ε, περιμένουμε να έρθει. Αρχίσαμε λίγο νωρίτερα. Και η επόμενη συμμετέχουσα στο πάνελ έχει και ένα, ε, μια πολύ σημαντική σύσκεψη που θα πρέπει να αρχίσει νωρίτερα, οπότε θα μας μιλήσει εκείνη πρώτη. Ε, σας καλωσορίζουμε κυρία Έκα και Σελασβίλη. Ε, πρώην Υπουργό παρά τον Πρωθυπουργό και Υπουργό Εξωτερικών ε, της ε, Γεωργίας. Τώρα, αυτή τη στιγμή, είσαστε πρόεδρος του Γεωργιανού Ινστιτούτου για στρατηγικέ Στρατηγικές Μελέτες. Είστε ειδικό σε θέματα ασφάλειας στην περιοχή αυτή. Έχετε, λοιπόν, το λόγο. Χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση, οι χώρες περιοχής ε, πάντοτε μας ανησυχούν όταν ακούμε να γίνονται ε, ασκήσεις στον Κάφκασο. Όπως έγινε μια άσκηση και πριν ξεσπάσει ο πόλεμος στη Γεωργία και τώρα Μας ανησυχεί ο χώρος στον οποίο γίνονται οι ασκήσεις. Ε. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ που είσαστε όλοι εδώ και θέλετε να μάθετε για το τι γίνεται ε, γενικότερα στο στρατηγικό περιβάλλον για το, το, το ανατολικό τμήμα της Ευρώπης και για την άσκηση αυτή. Ε, φυσικά αυτό εντάσσεται στο γενικότερο μοσαϊκό της κατάστασης ως προς την ασφάλεια που επικρατεί στην περιοχή. Για τις λεπτομέρειες ε, ο πρέσβης ε, θα σας κάνει μια λεπτομερή τεχνική στρατιωτική παρουσίαση. και κανονικά μετά από αυτή την ε, διεξοδική παρουσίαση της στρατιωτική πτυχή θα έπαιρνα κανονικά το λόγο, αλλά τώρα αντιστράφηκε η σειρά για να... Θα εγγραφεί όμως δεν πειράζει αυτή η τεχνική παρουσίαση σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Ε, πώς έγινε ο σχεδιασμός ε, σε ποιο μέτρο έχει εφαρμοστεί, ε, γιατί μιλάμε για την ενότια περιοχή της, ε, του στρατιωτικού μηχανισμού της Ρωσικής Ομοσπονδίας και για τη συγκεκριμένη στρατιωτική άσκηση και θέλω να δούμε ποιο είναι το μοντέλο που ακολουθείται με συστηματικό τρόπο και ποιος μπορεί να είναι ο στόχος μιας τέτοιας άσκησης, τέτοιας κλίμακας και με συστημικό τρόπο εφαρμόζεται από τη Ρωσία. Είπε η Πρόεδρος πως ήδη αυτή είναι μια πρώτη ένδειξη του μοντέλου που ίσως ε, άρχισε να ακολουθείται το 2008 ε, μετά την εισβολή και Μπορούμε να πάμε ακόμη και πίσω στο 2007 με τον ε, Σέρτζικοφ, τον Υπουργό Άμυνας για τον εξυγχρονισμό, αύξηση δαπανών για τον εξυγχρονισμό της ε, στρατιωτικής υποδομής ε, και όχι μόνο αύξηση αμυντικών δαπανών για τα στρατιωτικά παιχνίδια, αλλά και ε, για την συστηματοποίηση του μοντέλου για τις ε, και σχεδιαζόμενες ή ε, ευνίδιες ασκήσεις που ε, δρομολογεί με συστηματικό τρόπο πλέον η Ρωσία. Το 2008 στον Κάφκασο ήταν διαφορετικά τα δεδομένα, διότι ξαναλέω τότε γεννήθηκε αυτό το νέο μοντέλο και το 2014 είδαμε κάτι που υποτιμάται συχνά. Πριν από την προσάρτηση της Κρυμαίας έγιναν στρατιωτικές ασκήσεις εκεί και ε, είδαμε τα σενάρια των ενόπλων δυνάμεων που χρησιμοποιήθηκαν και στη συνέχεια για να γίνει η προσάρτηση της Κρυμαίας. Ε, πριν περάσουν δηλαδή σε, στο μάχημο κομμάτι είχαν γίνει οι ασκήσεις πριν γίνει η προσάρτηση, πριν γίνει η εισβολή. Ε, για να κάνω μια σύνοψη. Εκπαιδεύονται οι ένοπλες δυνάμεις από τη Ρωσία για ε, περιφερειακή αμυντικές θετικού τύπου επιχειρήσεις. Δεν πρόκειται για αμυντικές επιχειρήσεις, δεν εκπαιδεύονται για αυτό. Ε, πρόκειται για μάχημες ομάδες από όλα τα όπλα που εκπαιδεύονται με τρόπο ώστε να μπορέσει να σχεδιάσει η Ρωσία τους περιφερειακούς πολέμους όπου μπορούμε να έχουμε επιχειρησιακούς πυρήνες, ε, έναν ή πολλαπλούς. Ε, πρόκειται για σοβαρό εξοπλισμό λοιπόν, που εμπλέκεται σε αυτές τις ασκήσεις. Επίσης, στρατηγικό και τακτικό σχεδιασμό διαφορετικών τακτικών μαχήμων ομάδων, ούτω ώστε ε, να ε, εμπλακούν σε εξορισμού περιφερειακές επιχειρήσεις και είδαμε ότι η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτές τις ομάδες προσδίζοντα ένα στρατιωτικό σκέλος αυτές τις ασκήσεις Είδαμε επίσης ότι αυτό σχετίζεται όχι μόνο με το νότο της Ρωσικής Ομοσπονδίας αλλά και με την Ανατολή και ε, ε, Δύση, ε, μπλέκονται και με μέλη του ΝΑΤΟ και όταν μιλάμε για τον νότο ε, της Ρωσικής Ομοσπονδίας εξυπακούεται ότι εμπλέκεται το ανατολικό ε, κομμάτι της Ευρώπης, ε, πόντος, ε, αλλά πρόκειται και για χώρες φυσικά όπως η Ουκρανία και η Γεωργία. Επιδεινώνεται λοιπόν το περιβάλλον της ασφάλειας και έχουν και συμβολικό χαρακτήρα αυτές οι ασκήσεις, ε, όχι μόνο πρακτική σημασία, Θέλει να δείξει ότι έχει εξυγχρονισμένες ένοπλες ε, δυνάμεις που μπορεί να χρησιμοποιήσει ούτω ώστε να, ε, να είναι σε εγρήγορση και να μπορούν ε, να είναι σε ετοιμότητα και να αναπτυχθούν ταχύτατα. Υπάρχουν ε, οι κανονικές ε, επιχειρήσεις, Κάφκασος 2016, σχεδιασμένη επίθεση μεγάλης, πάρα πολύ μεγάλης ε, εμβέλειας και κλίμακας και βλέκεται και ο θολίσκος της Κασπίας. Ε, για γεωπολιτικούς λόγους οι ευνίδιες ασκήσεις είναι που είναι σημαντικές διότι εξασφαλίζουν ότι οι ομάδες μπορούν να εμπλακούν σε επιχειρήσεις ε, αμελητή. Σε ευνίδιες ασκήσεις προσπαθεί να εξασφαλίσει η Ρωσία ότι οι επιχειρήσεις όχι μόνο στον Νότο αλλά γενικότερα ε, ε, είναι σε ετοιμότητα και μπορούν να αναπτυχθούν το ταχύτερο δυνατόν. Οπότε πάνω ε, από το 75% της ετοιμότητας έχει επιτευχθεί και μπορούν να περάσουν ε, σε μάχημη κατάσταση αν χρειαστεί. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ο πολιτικός πόσο είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό διότι μπορεί η Ρωσική Ομοσπονδία να αποφασίσει να εμπλακεί σε συγκρούσεις πέρα από τις γειτονικές χώρες και πρέπει να είναι σε ετοιμότητα και ξαναλέω χάρη σε αυτές τις ευνηδιαστικές ε, επιθέσεις που είναι ε, απρόβλεπτες αλλά δυστυχώς λένε και πιο συχνές επιτρέπουν αυτή την ετοιμότητα. Τις έχουμε παρατηρήσει στον Κάφκασο και ε, συχνά βλέπουμε ότι ε, επηρεάζονται χώρες εντός και εκτός ε, του ΝΑΤΟ, δηλαδή υπάρχει αυτό το μοντέλο προσπαθεί ε, να καταστήλει τις δικές μας προσπάθειες εντός ή εκτός του ΝΑΤΟ να έχουμε περιφερειακές πλατφόρμες Αζερβαϊτζάν, Τουρκία, Γεωργία για συνεργασία της Ένωσης με άλλες χώρες. Και όταν μιλάμε για το μοντέλο για, τη, το περιβάλλον ασφάλειας που επιδεινώνεται γύρω από τις ε, γειτονικές ε, της Ρωσίας χώρες, ε, πρόκειται για ικανότητες α2AD. Ε ε, βλέπουμε λοιπόν το μοντέλο όχι μόνο στα δυτικά της Δοσκής Ομοσπονδίας Βαλτικές χώρες, αλλά και στον Εύξηνο Πόντο. Ε, προσάρτηση της Κρυμαίας. Μπόρεσε η Ρωσία να διευρύνει την κλίμακα και την ένταση του στρατιωτικού εξοπλισμού που υπάρχει επιτόπου ούτως ώστε οι χώρες του ΝΑΤΟ να μην μπορέσουν να ε, τόσο αποτελεσματικά να ε, οργανώσουν την άμυνά τους λόγω των δυναμικοτήτων, ε, των ικανοτήτων, συγγνώμη, AD που βρίσκονται επί τόπου. Ε, και όταν μιλάμε για τη Νότια Οσετία, για τη Γεωργία, πέρα από τον Κάφκασο διαπιστώνουμε ότι ακόμη και για τους πυράβλους, ε, εδάφους, αερά, για τα Ισκάντερ, για τα... Ε, έχουν εμβέλεια 500 χιλιόμετρα, οπότε είναι ξεκάθαρα οι ικανότητες AD. Ρωσία θέλει να έχει μια πλήρη έννοια ε, για την παρουσία στρατιωτικής βάσης. Μέχρι στιγμής αυτό έχει υλοποιηθεί μόνο στην Αρμενία. Ε, κανείς δεν έχει ε, ψευδεστήσεις για τη στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας ε, φυσικά υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους συμβαίνουν αυτά στη γειτονική μας χώρα, αλλά εξακολουθεί να ισχύει αυτή η κατάσταση ε, στο Διούμρι και στην αεροπορική βάση έξω από το Γέρεβανος έχει πάρει ε, η Ρωσία την άδεια εδώ 45 χρόνια και αναπτύσσει τον στρατιωτικό εξοπλισμό σε αυτές τις δύο βάσεις ε, και χρησιμοποιήθηκαν και για τις επιχειρήσεις ε, στη Συρία. Οπότε ε, ο Κάφκας δεν έχει μόνο σημασία σε σχέση με την παρουσία της Ρωσίας σε στρατιωτικές επιχειρήσεις στην Ανατολική Ευρώπη στον Εύσκηνο πόδο. Όχι, συνδέεται με τον τρόπο που αντιλαμβάνεται τη παρουσία της στη Ρωσία και στη Μέση Ανατολή η Ρωσία. Οπότε υπάρχει υπάρχουν διαφορετικά συμφέροντα και ενίοτε εστίαση στα συμφέροντα της Μέσης Ανατολής. Ε, βλέπουμε ε, την Ρωσία να ρευσπαστικοποιείται, ε, κυρίως στη Ρωσία. Δηλαδή αυτά που συμβαίνουν στο Κάφκασο έχουν σημασία σε σχέση και με τους στόχους της Ρωσικής Ομοσπονδίας ε, στη Μέση Ανατολή. Για να μην μακρηγορώ, για να μην μονολογώ και για να αξιοποιήσω αποτελεσματικά τον πολύτιμο χρόνο που έχουμε. Θα κλείσω εδώ και θα είμαι στη διάθεσή σας για να απαντήσω σε τυχόν ερωτήσεις. Εν είδη σύνοψης, μία πρόταση είναι ανησυχητικό ο τρόπος με τον οποίο αλλάζει το περιβάλλον ασφαλείας, και φυσικά η προσάρτηση της Κρυμαίας ε, άλλαξε τη διάσταση του προβλήματος και τις στάσεις ε, της Ρωσίας για αυτά τα ζητήματα με πολύ ανησυχητικό τρόπο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ για την πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η εισαγωγή. Καλωσορίζω τώρα τον επόμενο μιλητή που είναι ο Ασκόν Χρέη Προϊσταμένου της Αποστολής της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ ο πρέσβης Ιγκόρ Μπόσχοκ. Δεν ξέρω αν πρόφερα σωστά το όνομά σας. Ευχαριστώ πάντως. Μπορείτε να μας παρουσιάσετε τις στρατιωτικές πτυχές. Τη στρατιωτική άσκηση Κάφκασο 2016. Εν συνεχεία θα περάσουμε στη συζήτηση. Λοιπόν, ακούμε την παρουσίαση, καταρχήν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Τιμή και χαρά που είμαι εδώ. Είναι πολύ σημαντικό για μένα και σας ευχαριστώ που συγκαλέσατε αυτή τη συνεδρίαση για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα, για να μιλήσουμε λιγάκι για το τι συμβαίνει μέσα και γύρω από την Ουκρανία, στα πλαίσια όχι μόνο της ασφάλειας Ουκρανίας, αλλά της περιφερειακής και παγκόσμιας ασφάλειας. Γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό τώρα. Το σημαν... Λέγομαι Ιγόρο Μποζόκ. Είπατε την ιδιότητά μου. Ασχολούμαστε με θέματα όπως αυτό που μας απασχολεί σήμερα σε καθημερινή βάση με τους συναδέλφους και εταίρους στο ΝΑΤΟ. Υπάρχει μια αμφίδρομη δράση, δίνουμε και παίρνουμε πληροφορίες. Ο στόχος είναι να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε όχι μόνο τις, στρατηγικές, αλλά και στρατηγικές και παγκόσμιες προοπτικές των επιθετικών τάσεων της Ρωσίας που επανεκκίνησαν είχαν πρώτη φορά ξεκινήσει το 2014. Λοιπόν, το θέμα μας είναι ο Κάφκασος 2016. Είναι πολύ σημαντικό αυτό το θέμα, αλλά είναι μόνο μία ψηφίδα από μία γενικότερη στρατηγική της Ρωσικής Ομοσπονδίας που σκοπό έχει να αποκαταστήσει τη γεωπολιτική της Σοβιετικής Ένωσης. Ο στόχος της Ρωσική Ομοσπονδία και όλων των δραστηριοτήτων της είναι όχι η Ουκρανία, δεν ήταν η Γεωργία, δεν ήταν η Υπερνηστερία, ούτε η Αφχασία, η, η Νότια Καυκασία, ούτε το Καραμπάχ, αλλά η αποκατάσταση που, αυτού που είπε ο Πούτιν κατ' επανάληψη η μεγάλη, που ονόμασε η μεγαλύτερη απόλυτη του 20ου αιώνα, η κατάρρευση δηλαδή, της ε, Σοβιετικής Ένωσης, της ΕΔ και των δορυφόρων της. Η άσκηση ΚΑΦΚΟΣ 2016 είναι τμήμα ενός ευρύτερου μοσαϊκού που προσπαθεί να δημιουργήσει το Κρεμλίνο για να ενισχύσει τη στρατιωτική του δύναμη. Να έρθει πιο κοντά στις ε, κρίσιμες στρατιωτικά περιοχές της ε, σφαίρας του, τόσο ώστε να επιδεινώσει τη θέση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, καθώς και των συμμάχων τους. Εμείς δεν πιστεύαμε το 2008 ότι η άσκηση του Κάφκασου ήταν η προετοιμασία μιας γενικότερης δράσης. Κάτι κάποιου πράγματος το οποίο θα κατέληγε δηλαδή σε εισβολή ή σε απόπειρα εισβολή της Γεωργίας. Αυτή τη φορά βλέπουμε τα σημάδια, τους προδρόμους α, παρόμοιων προετοιμασιών, παρόμοιων προσπαθειών. Και γιατί το λέω αυτό. Αν μιλάμε για τις κινήσεις της Ρωσικής Ομοσπονδίας και των δυνάμεών της όλο και πιο κοντά στα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ζητώ συγγνώμη, μπερδέθηκα με το μικρόφωνο, γιατί είναι η πρώτη φορά που χρησιμοποιώ τέτοιο μικρόφωνο. Και μπερδέθηκα και με, τον, με το PowerPoint. Αν μιλάμε για την ε, σφαιρική εικόνα, είμαι υποχρεωμένος να επανέλθω στην ε, Ανατολική Ουκρανία. Γιατί στις 15 Σεπτεμβρίου φέτος η κατάπαυση του πυρός ήταν κάτι που είχε αναγγελθεί. Η επόμενη, η μειωστή ε, κατάπαυση του πυρός είχε αναγγελθεί, η οποία όμως ήταν λιγάκι διαφορετική. Γιατί και οι στρατιωτικοί συμμετείχαν, ε, συμμετείχαν και, και ε, συμφωνήσαν με αυτή την κατάπαυση του πυρός. Μειώθηκαν ο αριθμός ε, των όλμων, των βολών κτλ. Συνεχίστηκαν όμως οι βολές. Την τελευταία εβδομάδα είχαμε περίπου 30 βομβαρδισμούς τη μέρα. Χθες είχαμε 15 περίπου βομβαρδισμούς τη μέρα. Αλλά συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί και ο στόχος είναι να προκαλέσουν να προκαλέσουν τους Ουκρανούς στρατιωτικούς που προστατεύουν ε, την περιοχή για να αντιδράσουν ούτως ώστε να εξαπολύσουν στρατιωτική δράση για να διεισδύσουν περαιτέρω στο έδαφος της Ουκρανίας ή να αποκαταστήσουν τη χώρα μας εν το συνόλο της. Δεν βομβαρδίζουν τώρα με όπλα τα οποία απαγορεύει η Συμφωνία Μίσκ, αλλά ε, με μικρά όπλα. Ε, μερικές φορές ρίχνουν και χειροβομβίδες, RPG και τα λοιπά. Λυπούμε που τα λέω όλα αυτά, γιατί θυμάμαι πότε ξεκίνησε. Ε, ο πρώτος βαρδισμός ήταν σκάνδαλο. Τώρα μιλάμε για 14-15 βομβαρδισμούς και αυτό θεωρείται επιτυχία. Αλλά ταυτόχρονα καταστρέφεται το έδαφος, η υποδομή. Ε, προκαλούνται τραυματισμοί και ε, των το στρατιωτών μας και πεθαίνουν στρατιώτες μας. Ελπίζω όμως ότι αυτή η τάση μείωση των βομβαρδισμών τελικά θα οδηγήσει σε μια διαρκή κατάπαυση του πυρός, ούτως ώστε να ανοίξει το πολιτικό μονοπάτι για να επιληθεί η κρίση αυτή στην Ουκρανία προκάλεσε η Ρωσία. Αλλά έχουμε κάνει μια ανάλυση και δεν επιβεβαιώνει κάτι τέτοιο. Γιατί? Γιατί παράλληλα με τους βομβαρδισμούς η Ρωσία ε, στήριξε τους στρατιωτικούς στην Ανατολική Ουκρανία και δεν απέσυρε τα όπλα της ε, από τα σημεία αποθήκευσης με βάση τα όσα προβλέπει η Συμφωνία Μίσκ, ε, με βάση τους υπολογισμού μας. Αυτή η αποχώρηση των οπλισμών από τη Ρωσία και από του στρατιωτικού που στήριζε στην Ανατολική Ουκρανία η Ρωσία ολοκληρώθηκε μόνο κατά 35%. Έχει περάσει ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και αυτό αποδεικνύει ότι δεν έχουν καμία τέτοια πρόθεση στην πραγματικότητα να αποσύρουν τον οπλισμό τους και να πετύχουμε μία πραγματική και βιώσιμη κατάπαυση του πυρός. Παράλληλα, η Ρωσία έχει ε, μια ισχυρή στρατιωτική παρουσία ε, στα ανατολικά και βόρεια σύνορα με την Ουκρανία. Είναι πολύ επικίνδυνο αυτό γιατί αυτή η στατιωτική παρουσία έχει 440 μαχητικά αεροπλάνα και καμία τρακοσαριά ε, μαχητικά ελικόπτερα για να υποστηρίξει χερσαίες επιχειρήσεις για να μπορέσει να διευρύσει περαιτέρω το έδαφος της Ουκρανίας. Ε, η στρατιωτική παρουσία, ε, η παρουσία που στηρίζει στην Ανατολική Ουκρανία είναι, βασίζεται σε 41.000 στρατιώτες που συμπεριλαμβάνει 6.000 τακτικά ε, τακτικές μονάδες στρατιωτών από τη Ρωσία. Και εδώ σας μιλάω μόνο για την ανατολική α, Ουκρανία, θα μιλήσω μετά για την Κρυμαία. Αυτή η στρατιωτική παρουσία της Ρωσίας εντός της α, ε, Ουκρανίας σημαίνει 600 τάγκ μάχης. Μπορώ να σας απαριθμίσω πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και συμμάχους του ΝΑΤΟ που έχουν πολύ λιγότερα τάξ στο τακτικό του στρατό. από αυτά τα ρωσικά τάγκ. Δεν θα σας μιλήσω για τα υπόλοιπα όπλα ε, και δεν θα σας δώσω νούμερα. Είναι πάρα πολλά. Η Ρωσία επίσης εξακολουθεί να εφοδιάζει και να τροφοδοτεί αυτά τα παραστριωτικά, τις παραστριωτικές ομάδες με πυρομαχικά, επιμελητεία, εξοπλισμό. Γιατί. Το ερώτημά μου είναι γιατί. Το συμπέρασμά μας είναι ότι ο στρατηγικός στόχος της Ρωσίας παραμένει ο ίδιος. Να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο της Ουκρανίας και να δημιουργήσει έναν πραγματικό στρατό για να καταστρέψει εντελώς το περιβάλλον ασφαλείας στην περιοχή, απειλώντας περαιτέρω την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον ΝΑΤΟ και τους συμμάχους τους. Και να αποκαταστήσει βάθμιδόν την σοβιετική γεωπολιτική αρχιτεκτονική στην περιοχή αυτή. Για να το κάνει αυτό, για να το καταφέρει αυτό, για να το επανεκκινήσει μετά τη Ρωσία, ε, οι Ρώσοι εισέβαλαν και προσάρτησαν την Κρυμαία από την Ουκρανία. Προσπάθησαν να το παρουσιάσουν ως μια συμβολική κίνηση, την αποκατάσταση της ιστορικής αλήθειας, ότι υλοποιούν τη θέληση του πληθυσμού επιτόπου, αλλά η στρατιωτική του στόχη και η ε, στρατηγική του στόχη ήταν εντελώς διαφορετική. Χρειάζονταν τέτοια όπλα για να εξασφαλίσουν ότι θα υπάρξει ε, στρατιωτική ε, παρουσία για να αποσταθεροποιήσουν την Ευρωπαϊκή Περιοχή, την Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τους συμμάχους που προσπαθούσαν να βοηθήσουν την Ουκρανία για να κρατήσουμε σε καλή κατάσταση την ασφάλεια. Ε, η Κρυμαία θεωρείται τεράστιας γεωστρατηγικής σημασίας από το Κρεμλίνο. Ο βασικός στόχος της Ρωσίας στην Μαύρη Θάλασσα είναι Θα σας μιλήσω για αυτά που βλέπετε εδώ, που είναι εντυπωσιακά νούμερα. Είναι να εξασφαλίσει τις προϋποθέσεις ώστε να παρεμποδίσει την επανένωση Ουκρανίας Κρυμαίας. Αυτό είναι ένας μικρός ε, τακτικός στόχος και να αποτρέψει την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και τις Ηνωμένες Πολιτείες ε, από το να αστυνοποιηθούν στον έξινο πόντο, να δημιουργήσει αντιστάθμισμα στην πρόσφατη πρωτοβουλία που ξεκίνησε με, τους, με τη βαλιστική αντιπυραυλική άμυνα ε, που εγκαταστάθηκε στη Ρουμανία, ε, να μην υπάρξει κάτι τέτοιο, μια αντίστοιχη αμυντική προσπάθεια στην Κρυμαία και στην ευρύτερη περιοχή θέλουν να συνεχίσουν τη διείστηση στην Μέση Ανατολή και να υπάρξει στρατιωτική παρουσία για να ενισχυθεί η ναυτική παρουσία της Ρωσικής Ομοσπονδίας στη Μεσόγειο. Για να υλοποιηθούν αυτοί οι στόχοι, οι Ρώσοι δεν χρειάζονται μόνο το, τη χερσόνησο της Κρυμαίας, χρειάζονται περισσότερα και μεγαλύτερα εδάφη. Γι' αυτό τώρα όμως ενισχύουν την Κρυμαία. Και τώρα θα δούμε τα νούμερα. Έχουμε στην Κρυμαία τώρα οι κοινέ ε, task force της Ρωσικής Ομοσπονδίας έχουν τακτικά στρατεύματα, τακτικές δυνάμεις. Δεν είναι κάποιοι αντάρτες, ε, δεν είναι άταχτα, άταχτες ε, μονάδες. Έχουμε 29.000 περίπου στρατιώτες και αν δείτε τα νούμερα στην οθόνη, όταν κατέρευσε η Σοβιετική Ένωση οι τακτικές δυνάμει στην Κρυμαία ήταν 70.000 στρατιώτες. Αργότερα, Ρωσία και Κρυμαία, τα νόμιμα στρατεύματα που ήταν παρόντα στην Κρυμαία ήταν 12.500. Τώρα μετά την παράνομη προσάρτηση της Κρυμαίας έχουμε φτάσει στις 29.000 και τα σχέδια είναι να φτάσουμε στις 43.000 ε, στρατιώτες ο πλευρά Ρωσίας. Θέλουν να αποκαταστήσουν δηλαδή την ισχύ των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων μέχρι να, κοινοθώσουν στο επίπεδο της Σοβιετικής εποχής. Η, η Σοβιετική Ένωση είχε στρατιωτική παρουσία στην Κρυμαία με σκοπό να αποτρέψει και να επιδεινώσει την κατάσταση των εχθρών, εν πάση περιπτώσει. Το ΝΑΤΟ, και τις δυτικές δυνάμεις. Έχουμε 600 τάγματα, ε, ε, συγγνώμη, μάχημα τάγκ, Να μην σας ε, κουράσω με νούμερα, γιατί το ή έχετε όλοι τις διαφανίες μου. Αυτή είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα εικόνα. Είναι η κατάσταση στην παράκτια ακτοφυλακή στην Χερσόνησο της Κρυμαίας. Έχουμε 15 χωριστές ε, ταξιαρχίες ε, που εδρεύουν στη Σεβαστούπολη. τι έχουν κινητά πυραυλικά συστήματα με βεληνικές 320 ε, χιλιόμετρα και δυνατότητα ε, πλήγματος 420 χιλιόμετρα. Βλέπετε τον μπλε κύκλο πάνω στην οθόνη. Εδώ η πύραυλη της Ρωσίας βλέπετε ότι μπορεί να φτάσουν γρήγορα στην, σε χερσαία εδάφη και οι πύραυλοι μπορούν να πλήξουν επίσης και ναυτικούς στόχους. Εάν μου πείτε ότι αυτό είναι αμυντική προσπάθεια, αμυντικές δυνάμεις, το αμφισβητώ. Αυτό έχω να σας πω. Όπως σας είπα λοιπόν, ο στόχος είναι να ενισχύσουν και να δημιουργήσουν ένα στρατό ένα στρατό λοιπόν να δημιουργήσουν, τόσο ώστε να εξασφαλίσουν ένα στρατιωτικό δυναμικό επίθεσης των παράκτιων ε, κρατών της ε, Μαύρης Θάλασσας, δηλαδή τους μη συμμάχους της ε, Ρωσικής Ομοσπονδίας, και κανένα δεν σύμμαχο δεν έχει αυτή τη στιγμή, και να δημιουργήσει ένα στρατό ούτω ώστε να επεκτείνει το στρατιωτικό της δυναμικό πέραν του εύξηνου πόντου και να αποτρέψει τις προσπάθειες ε, των, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των συμμάχων να δημιουργήσει τις συνθήκες για να αποκτήσει τον πλήρη έλεγχο στον εύξηνο πόντο. Αυτός είναι ο γενικός στόχος. Ο μικρότερος στόχος είναι να δημιουργήσει ένα στρατό, ούτως ώστε να προετοιμάσει πιθανές στρατιωτικές επιχειρήσεις διείσδυσης στην Ουκρανία από νότου. από τον Νότο. Από τη Χερσόνησο της Κρυμαίας θα προσπαθήσει να πάει προς την υπηρετική Κρυμαία, είτε χερσαίος, είτε έμεσα, παραθαλάσσια, μέσω της του, του κόλπου της Χερσόνησου της Οδυσσού. Και για να, το, να, τσεκάρει το δυναμικό αυτό συγκέντρωσης ε, δυνάμεων στην Κρυμαία για να ετοιμαστεί λοιπόν, εάν ληφθεί η απόφαση του Κρεμλίνου, η άσκηση αυτή Κάφκασος 2016 έλαβε χώρα πολύ κοντά στα Ουκρανικά σύνορα. Ένας από τους στόχους ή μάλλον από τα σενάρια. Πριν περάσουμε στα σενάρια όμως να σας πω κάτι άλλο. Είναι σημαντικό να κοιτάξουμε αυτή την εικόνα. Εδώ βλέπετε τις, α, τους μηχανισμούς έτσι, εξαπάτης που χρησιμοποιεί το Κρεμλίνο σε όλα τα διεθνα, διεθνή φόρουμ. Αυτή η άσκηση Κάφκασος 2016 είχε δύο δέσμες δεδομένων. Αυτά που δηλώθηκαν για το στρατιωτικό προσωπικό που συμμετείχε στην άσκηση. 12.000 λέει. Στην πραγματικότητα 100.000. Και τα όπλα ήταν διαφορετικά. Τάγκς και τεθωρακισμένα. 400 ε, δήλωσαν οι Ρώσοι. Στην πραγματικότητα 10.000. Μπορούμε να συνεχίσουμε με τα αριθμητικά στοιχεία. Δεν θα τα διαβάσω, τα βλέπετε στην οθόνη σας. Αυτό που είναι σημαντικό και ανησυχητικό για την Ουκρανία και ο λόγος που φοβηθήκαμε ήταν ο εξή. Θα ακούσατε ίσως ότι στην περιοχή που προσωρινά ε, κατέχει ε, η Ρωσία, στον Τονές και στο Λουχάνσκ, έχει δημιουργήσει δύο στρατιές. Ε, έχουμε τους μισθοφόρους και παραστρατιωτικούς, έτσι τους λένε, αλλά στην πραγματικότητα είναι τακτικές δυνάμεις ε, των νότιων ε, δυνάμεων της Ρωσίας που βρίσκονται στις προσωρινά κατεχόμενες αυτές σε περιοχές του Ντονέσκ και του Τουλουχάς. Και αυτές οι δυνάμεις της Ρωσίας συμμετείχαν στην άσκηση Κάφκασος 2016. Ήταν τμήμα αυτής της προσπάθειας. Και ένα από τα σενάρια είναι επίθεση πεζοναυτών στην παράκτια περιοχή του εχθρού. Αυτό μας φόβησε πάρα πολύ. Αυτό το σενάριο. Γιατί τον έχεις 12.000 στην Κρυμαία μαζί με 41.000 στρατιώτες στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας, στο εσωτερικό ε, των περιοχών Ντονέσκ και Λουχάνσκ, φτάνουμε περίπου στις 70.000 στρατιώτες. 70.000 στρατιώτες που μπορεί να είναι σε θέση να επιτεθούν. Εμείς είμαστε έτοιμοι να αντισταθούμε φυσικά, Παρακτηρήσαμε τις κινήσεις, προσπαθήσαμε να τις αναλύσουμε, να κυκλοφορήσουμε τις πληροφορίες και να προετοιμαστούμε. Παράλληλα, αυτή η οικοδόμηση, αυτή η αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας δεν είναι η τελική, δεν είναι ο στόχος αυτός. Είναι ένα από τα βήματα των Ρώσων προς το ευρύτερο, το μεγαλύτερο στόχο. Και για να σταματήσουμε αυτή την προσπάθεια θα πρέπει όλοι να πιέσουμε την ε, Ρωσική Ομοσπονδία και την κυβέρνησή τη, θα πρέπει να ασκήσουμε από κοινού προσπάθειες για να αναγκάσουμε το Κρεμλίνο να σταματήσει αυτή την επιθετική ε, πολιτική και αυτή την ε, αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας τους. Γιατί όπως σας είπα αυτή η αύξηση της στρατιωτικής παρουσίας της Ρωσίας δεν είναι μόνο κατά της Ουκρανίας, είναι τμήμα μιας μεγαλύτερης στρατηγικής και δεν στρέφεται μόνο εναντίον μας, της Ουκρανίας δηλαδή, αλλά εναντίον όλων μας. Πώς θα τους αναχαιτήσουμε, την απάντηση την ξέρουμε. Με πολιτική πίεση και κυρώσεις. Γι' αυτό είναι σημαντικές οι κυρώσεις. Φυσικά όλοι καταλαβαίνουμε ότι είναι πολύ καλή και πολύ ελκυστική η ρωσική αγορά. Επίσης, καλά είναι τα λεφτάκια τους, τα, ρούβια, τα τους, αλλά Είμαστε έτοιμοι να ξεπουληθούμε, να ξεπουλήσουμε τη σταθερότητα και την ασφάλειά μας σε όλη την περιοχή. Και ό,τι έχει οικοδομηθεί μετά την ε, κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης. Πρέπει να απαντήσουμε σε αυτό το ερώτημα. Σας ευχαριστώ. Ambassador, thank Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρέσβη, για την παρουσίαση αυτή. Ακούσαμε μια φωνή από την περιοχή την, με την οποία και συμφωνώ. Ασφαλώς όταν μιλούμε για την κοινή πρόσληψη απειλών είναι εξαιρετικά σημαντικό να έχουμε συνείδηση των πραγματικών στοιχείων για τη συνεδρίαση αυτή. Ο κύριος Γκάλερ. Ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή και την επισκόπηση που λάβαμε. Η πολιτική μας θέση πρέπει να παραμείνει ως έχει. Γι' αυτό και θα έλεγα ας παραμείνουμε ενωμένοι στην προσέγγιση μας προς τη συνεχιζόμενη επιθετικότητα και ας μεταφέρουμε το μήνυμά μας μέσω των διάφορων διάβλων διαλόγου που υπάρχουν αλλά όπως βλέπουμε επίσης όσον αφορά τη Συρία όπου η Ρωσία δραστηριοποιείται από την πλευρά του καθεστώτος Ασάντ και πομβαρδίζει ανηλαιώς την το Ανατολικό Χαλέπι με όλους τους άμαχους εκεί. Αυτό δείχνει μια αποφασιστικότητα να μην λαμβάνει η Ρωσία κανέναν υπόψη. Δεν βλέπουμε κάποιο ίχνος ότι θέλει να αλλάξει τη στάση της ή να επιστρέψει σε μια πολιτική σύμφωνη με το διεθνές δίκαιο. Γι' αυτό και η ερώτησή μου είναι, αν κοιτάξετε τους αριθμούς που μπορούν να τους αριθμούς των στρατευμάτων που μπορούν να κινητοποιηθούν. Δεν έχουμε να κάνουμε με εκπαίδευση, έχουμε πραγματικούς βομβαρδισμούς, έχουμε κατανάλωση εξοπλισμών και όλα τα σχετικά. Έχετε κάποιους αριθμούς ή εκτιμήσεις για το πόσο χρονικό διάστημα θα μπορούσαν να συνεχίσουν τέτοιες δραστηριότητες στη, στη Συρία, στην Κρυμαία και να διατηρήσουν τον εφοδιασμό των αντικαθ... αυτών που τους αντικαθιστούν στην Ανατολική Ουκρανία και στην Γεωργία. Είδαμε κάποια στρατόπεδα, προχειρά στρατόπεδα που έχουν εγκαταστήσει και στην Νότια Οσετία επίσης μια φορά το χρόνο έχουμε πλήρη εκπαίδευση Έχουμε κάποια γνώση του πόσο χρονικό διάστημα μπορούν να συνεχίσουν με αυτό. Επειδή αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι αυτή η παρατεταμένη παρουσία σε παράνομα κατηλημένες περιοχές συν τον επίκαιρο θερμό πόλεμο στη Συρία. Ποιες είναι οι εκτιμήσεις σας σχετικά με την Ουκρανία και την Γεωργία. Ευχαριστώ. Τον Πόσο Μαρακιούρεκ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρέσβη, ο πρόεδρος Ποροσέγκο απευθύνθηκε πριν από πολλούς μήνες σχετικά με την λεγόμενη αποστολή υλοποίησης των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ανατολική Ουκρανία. Η υλοποίηση σήμαινε πως με αυτόν τον τρόπο επρόκειτο να παρακολουθηθεί η συμφωνία του Μίνσκ, η εκεχηρία κτλ. Πιο πριν υπήρξαν επίσης προτάσεις για μια αστυνομική αποστολή, όπως και να έχει μια παρουσία των χωρών μας. Θέλω να ρωτήσω ποιες αντιδράσεις προκάλεσαν οι προτάσεις αυτές και σε ποιο βαθμό το ζήτημα είναι επίκαιρο για την Ουκρανία. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μία ερώτηση στους διακεκριμένους ομιλητές μας. Ακά μιλήσατε για ασκήσεις σκοπευτών ε, για ξαφνικές ασκήσεις που γίνονται παράλληλα με τις τακτικές από ό,τι ξέρω αυτό είναι κάτι καινούριο. Είναι ένας νέος τρόπος γρήγορης ετοιμασίας, γρήγορης στράτευσης. Ποια είναι η ιστορία τέτοιων ασκήσεων. Έχετε παραδείγματα στο παρελθόν τα οποία μπορείτε να μας παρουσιάσετε για μια στρατολόγηση αυτού του τύπου. Βλέπω ακόμα κάποιος ζητάει, ζητεί το λόγο, είστε σε ένα νέο κύκλο. Παρακαλώ, έχετε τον λόγο, ο κύριος Πρέσβης πρώτα. Στη συνέχεια η κυρία Βίλη Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος αλλά παραστατικός. Για πόσο χρονικό διαστήμα, κυρία Πρόεδρε. Βλέπουμε τα προβλήματα είναι εκεί. Δεν θα μάθουμε την αλήθεια. Φυσικά, ποτέ. Θα θολώνουν τα νερά, θα λένε είμαστε εντάξει. Αντικειμενικές ενδείξεις υπάρχουν όμως. Έχουν παγώσει συντάξεις και μισθούς άρχισαν να χρησιμοποιούν αποθεματικά ταμείων. Ε, επίσημες εκτιμήσεις υποστηρίζουν πως μέχρι το 2017 θα ξεμείνουν από πόρους και θα χρειαστεί να χρησιμοποιήσουν ένα λεγόμενο στρατηγικό ταμείο ή όπως ακριβώς λέγεται. Αυτό αφενός. Αφετέρου, είμαι 100% σίγουρος πως η επίκαιρη ρωσική διοίκηση δεν θα παραλάβει το σφάλμα του τελευταίου γέννη της Σοβιετικής Ένωσης. Δεν θα επιτρέψει ποτέ να επέλθει μια κατάσταση στην οποία δεν θα έχουν χρήματα. Με άλλα λόγια, δεν θα παίξουν τα πάντα. Μόνο έως ένα συγκεκριμένο όριο. Τώρα το πού είναι το όριο αυτό είναι δύσκολο να υποθεί. Αλλά υπάρχουν ενδείξεις ότι το όριο αυτό πλησιάζει. Οι κυρώσεις λειτουργούν. ήδη είναι υπερκαταπονημένοι. Έχουμε τη Γεωργία, την υπερδυστερία, τον Αγκόρνο Καραμπάχ, τη Συρία, την Ουκρανία, σε δύο σημεία. Όλα αυτά καταναλώνουν και πολύ μάλιστα. Και για την ισχύ και για τη συνέχιση του πόκερ αυτού με τη Δύση πρέπει να επενδύουν όλο και περισσότερο σε στρατιωτικές παραστάσεις Πιστέψτε με, εργάζομαι στον ΝΑΤΟ. Οι ασκήσεις κοστίζουν πολύ. Έχουν αποτελέσματα άλλο αυτό, αλλά σίγουρο είναι ότι κοστίζουν πολλά. Γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό να διατηρήσουμε αυτή την αλληλεγγύη. Ο στόχος αυτού για μένα είναι προφανής. Αυτή η επίσπευση διαφορετικών δραστηριοτήτων αποσκοπούν στη δημιουργία ψυχολογικής πίεσης προς τη Δύση, στο να πιστεί στο να πιστείτε να υποχωρήσετε. Γιατί. Επειδή οι κυρώσεις λειτουργούν. Αυτό είναι. Αυτό είναι το ζήτημα. Θυμάστε, από την αρχή υπήρξαν πολλές συζητήσεις κατά πόσον είναι μια εύλογη απάντηση, κατά πόσον η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρεται έξυπνα χρησιμοποιώντας τόσο μορφωμένα μέσα για να πείσει κανείς τον παραβάτη να επιστρέψει στις αρχές του διεθνούς δικαίου. Φυσικά ο στόχος του επιτιθέμενου ήταν να λάβει επίθεση ως απάντηση. Τώρα το ξέρουμε. Αλλά υπάρχουν όρια και οικονομικοί μηχανισμοί. για να επανέλθει στη λογική και στις αρχές δικαίου. Λειτουργούν ήδη. Φυσικά και είναι εύκολο να εξηγήσουμε στους ντόπιου πώς έχουμε έναν εχθρό και πώς πρέπει να πολεμήσουμε. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα χρόνια. Η Κρυμαία. Ακούσα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα από την ρωσική γκλουμπίνκα. Είναι πολύ μακριά. Είναι φωνές που υποστηρίζουν γιατί χρειαζόμαστε την Κρυμαία. Πού είναι αυτή η Χερσόνησος. Γιατί για να διατηρήσουμε το, την Χερσόνησο αυτή πρέπει να παγωθούν οι συντάξεις μας. Δεν έχουμε πάει ποτέ, ούτε πρόκειται να πάμε ποτέ. Πού είναι η λογική σε όλο αυτό. Και αυτές οι φωνές ήδη υπάρχουν. Προσπαθούν να τις καταστήλουν φυσικά. Αλλά οι δρόμοι είναι ενδιαφέροντας ενδιαφέρουν τα σημεία. Επειδή από εκεί αρχίζουν κάποιες φορές οι σεισμοί. Αυτή είναι η απάντησή μου για την ερώτησή σας. Η εκεχηρία, η αστυνομική αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παρεπιπτόντως ήταν πολύ εύκολο να καταλάβω τον συνομιλητή μου επειδή οι γλώσσες μας είναι πολύ παρόμοιες. Εκτός από κάποια πράγματα κατάλαβα σχεδόν τα πάντα. Όσον αφορά την υλοποίηση της αστυνομική αποστολή. δεν υπάρχει ακόμα συνένεση για μια τέτοια αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλοποίηση, η εφαρμογή της συμφωνίας του Μίνσκ απαιτεί την ομοφωνία όλων των μερών, αν και η Ρωσία αρνείται το ότι αποχωρεί από αυτή τη συμφωνία, αν και όλοι οι άλλοι βλέπουν ότι το κάνει οι αντικαταστάτες τους είναι πολλές φορές πολύ δημιουργικοί για την υπονόμευση και την οπισθοδρόμηση της διαδικασίας. Ίσως ακούσατε ήδη πως η ιδέα είναι πως αν έχουμε επί 7 μέρες με τέτοια βιώσιμη εγχειρία να αρχίσουμε με την αποχώρηση στρατευμάτων από την Ουκρανική πλευρά και από την πλευρά των μαχητών σε τρία βήματα, σε, τρία σημεία και να δημιουργήσουμε τετραγωνικές επιφάνειες τριών χιλιόμετρων χωρίς στρατιωτικές δυνάμεις όπου θα εισέλθουν παρατηρητές και ελπίζαμε πως μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου θα αρχίσουμε την ανάποδη, αντίστροφη μέτρηση για τη την αποχώρηση. Συνέβη κάτι όχι. Συνεχίζουν οι βομβαρδισμοί και ακόμα δεν μπορούμε να αρχίσουμε το πείραμα αυτό το οποίο υποστηρίζει η ρωσική πλευρά, το οποίο υποστηρίζουν οι μαχητές και όλοι και το οποίο ήταν ιδέα των φίλων μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα δούμε. Ακόμη ελπίζουμε, ελπίζουμε ειλικρινά. Πώς θα υλοποιηθεί, θα είναι τουλάχιστον η πρώτη ένδειξη. για μια εφαρμογή του λεγόμενου πολιτικού τμήματος της συμφωνίας του Μίνσκ και επειδή θέλουμε να το εφαρμόσουμε. Αλλά φυσικά χωρίς μια βιώσιμη εκεχηρία δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί με διεθνείς παρατηρητές. Το πράσινο φως θα δοθεί όταν οι δυνάμεις ασφαλείας του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης και άλλων διεθνών οργανισμών επιτρέψουν στους παρατηρητές τους να πάνε στην Ανατολική Ουκρανία. Αυτό θα είναι το πράσινο φως για εκλογές. Μετά από αυτό δεν θα υπάρχει καμία δικαιολογία πλέον για να, για να καθυστερήσει και άλλο το πολιτικό τμήμα της Συμφωνίας του Μίνσκ πιο πριν είναι πολύ δύσκολο. Και τις ξαφνικές ασκήσεις, οι ξαφνικές ασκήσεις, πιστεύω δηλαδή σαν το 2008, εκτός μικροφώνου, η άσκηση Κάφκαστος ανακοινώθηκε, αλλά με ένα μεγάλο ψέμα. Αντί για 12.000 συμμετέχουν 100.000 στρατιώτες, αλλά έχουμε πολύ συχνά ξαφνικές ασκήσεις στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας που περιγράφονται πολύ ζωντανά από τον διεθνή τύπο αλλά για μας ακόμα πιο σημαντικό είναι να επιστρέψουμε στην εμπειρία της γεωργίας. Να δούμε πώς χρησιμοποιήθηκαν οι ξαφνικές ασκήσεις για να πάρουν τα διδάγματα που έχουν σήμερα. Γι' αυτό δεν σας δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να συμπληρώσω κάποιες πτυχές που αναφέρθηκαν σχετικά με τις ξαφνικές ασκήσεις. Εάν κοιτάξουμε το πού βρίσκεται τώρα η Ρωσία όσον αφορά τους πολιτικούς στόχους και τις στρατιωτικές ικανότητές της και θα δούμε ότι πολλούς πόρους που επένδυσε η Ρωσία σε στρατιωτικό εξοπλισμό, σε ετοιμότητα πυρός και στην διαλειτουργικότητα των διαφορετικών στρατιωτικών σωμάτων της, οι οποίες συμμετέχουν από κοινού σε επιχειρήσεις μάχης, το οποίο κάνουν και μάλιστα μαζί με δυνητικούς τους σύμμαχους, ενδυναμώνοντας έτσι τις συμμαχίες που έχουν συνάψει. Παράλληλα, βλέπουμε μια μεγάλη πρόοδο της Ρωσίας, η οποία απαιτεί πόρους. και κατανοούμε πως υπό το επίκαιρο πολιτικό σύστημα με τις οικονομικές του διαστάσεις είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς πως μακροπρόθεσμα η ρωσική οικονομία θα μπορέσει να το διατηρήσει αλλά βραχυπρόθεσμα δεν έχουμε κάποια ένδειξη για το ότι θα σταματήσει αυτό πολύ γρήγορα. Έχουμε ένα δυναμικό αναμονής. Χρειαζόμαστε πιο πολύ ενεργά μέτρα. Αυτό σημαίνει την ενδυνάμωση της ανθεκτικότητας των χωρών στόχο. και ιδίως των στενών εταίρων των δύο οργανισμών. Όταν λέω ανθεκτικότητα εννοώ ένα ολοκληρωμένο πακέτο την πολιτική διάσταση της ανθεκτικότητας, δηλαδή την εδραίωση της δημοκρατίας, την οικονομική ανάπτυξη και παράλληλα ένα περιβάλλον ασφαλείας, το οποίο θα είναι ανθεκτικό στην απειλή που σημαίνει η Ρωσία για τις χώρες μας. Πιστεύω ακράδαντα πως τόσο στην Γεωργία όσο και στην Ουκρανία με το χρονοδιάγραμμα που έχουμε στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, ένας λόγος για τον οποίο βλέπουμε την Ουκρανία να επιβιώνει ως κυρίαρχο κράτος και να προ... προοδεύει στη δική της μεταρρύθμιση, είναι επειδή ο Ουκρανικός λαός αντιστέκεται στις ρωσικές ένοπλες δυνάμεις, την οποία αντίσταση δεν πίστευε κανείς πως υπάρχει, ούτε καν η Ρωσία. Βλέπουμε δηλαδή μια εδραίωση, εθελοντική εδραίωση και μια αύξηση των ικανοτήτων. Τον καθοριστικό ρόλο έπαιξε ωστόσο η αντίσταση της Ουκρανίας. Εμείς είχαμε μια πιο σύντομη εισβολή, αλλά αντισταθήκαμε όσο περισσότερο μπορέσαμε ώστε να προκληθεί μια διεθνής εμπλοκή η οποία σε κάποια στιγμή σταμάτησε αυτή την προέλαση και την καταστροφή των, της γεωργιανής κυριαρχίας. Ακόμη 20% του, των εδαφών μας βρίσκονται υποκατοχή. Και έχουμε χιλιάδες Ρώσους στρατιώτες στο μικρό μας κράτος. Έχουμε στρατιωτικές βάσεις τόσο στην Απχαζία όσο και στην Νότιο Οσετία. Έχουμε μεγάλο άψυχο και έμψυχο στρατιωτικό υλικό στη χώρα μας. Αλλά ως χώρα επιζήσαμε επειδή πολεμήσαμε για να επερασπιστούμε τη χώρα μας τόσο με τον πολιτικό τρόπο, ενδυναμώνοντας την ανθεκτικότητά μας και ταυτόχρονα ενισχύοντας τις ικανότητες αμυνάς μας. Υπάρχει ο συνδυασμός των δύο. Η μεταρρύθμιση των κρατικών μας θεσμών η ενίσχυση της οικονομίας, η ενσωμάτωση της γεωργίας στον οικονομικό χώρο της Ευρώπης. Έχουμε ένα ελεύθερο καθεστώς το οποίο μας αφήνει να σανόμαστε Ευρωπαίοι. Τόσο σε θεσμικό επίπεδο όσο σε επίπεδο ικανοτήτων έχουμε βασικά στοιχεία τα οποία μας επιτρέπουν να επιζούμε. Και αυτό είναι ένας συνδυασμός που δεν μας κάνει να αισθανόμαστε άνετα με την κατάσταση όπως είμαστε επειδή η κατάσταση επιδεινώνεται επειδή η Ρωσία αισθάνεται ότι υπερισχύει με τον εξοπλισμό της. Προσωπικά δεν το πιστεύω, αλλά είναι πεπισμένη πως είναι έτσι τα πράγματα, το οποίο σημαίνει ότι γίνονται πιο επιθετικοί. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι, να είμαστε ανθεκτικοί και να αντιστεκόμαστε. Παραδείγματο χάρη μέσω μεταρρυθμίσεων, μέσω όθηση στην οικονομία μας και η εμπειρία της γεωργίας δείχνει πως είναι εξαιρετικά δύσκολο αλλά όχι αδύνατο να ανοικοδομηθεί μια επιτυχής δημοκρατία ενώ μας σκοπεύει ένα όπλο. Δεν πρέπει να είμαστε υπερβολικά απεσιόδοξοι ή αισιόδοξοι για να επιζήσουμε. Το ζήτημα δεν είναι για πόσο χρονικό διάστημα μπορεί να επιβιώσει η Ρωσία, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε όσο αντέχει η Ρωσία. Δηλαδή πώς θα αναπτυχθούμε κατά τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος αυτού και πώς θα γίνουμε ανθεκτικοί έναντι της απειλής που σημαίνει η Ρωσία όσον αφορά την κατοχή τις περιοχές υπορωσική κατοχή και τις δράσεις της Ρωσίας επί εδάφους είναι αυτό που κάνει η Ρωσία στην Ανατολική Ρωσία. Προσπαθεί να διασφαλίσει πως η κατοχή θα αποτελέσει τμήμα μιας στρατιωτικής υποδομής της Ρωσίας. Ταυτόχρονα αποτελεί πολιτικό μηχανισμό μόχλευσης ενάντια των δημοκρατικά εκλεγμένων κυβερνήσεων στην Ουκρανία και στη Γεωργία. Γι' αυτό και αποτρεπόμαστε από το να επιλέξουμε εμεί πώς θα εξελιχθούμε ως κράτη, σε ποιες οικογένειες εθνών θα βρεθούμε στο μέλλον και πώς οι λαοί μας θα ασκήσουν τα κυριαρχικά τους δικαιώματα και θα είναι πολίτες ελεύθερων οικονομιών της αγοράς, ελεύθερων δημοκρατικών κρατών. Και αυτό γίνεται και στο μικρό επίπεδο της ανάπτυξης των χωρών μας. Όσον αφορά τις ξαφνικές ασκήσεις, Έχουμε τακτικές ασκήσεις μεγάλης κλίμακας με χρήση ολόκληρης της στρατιωτικής υποδομής αποτελούν έναν καλό τρόπο να ελέγξουν πώς θα μπορούσε να γίνει μια στρατιωτική επιχείρηση μεγάλης κλίμακας. Αλλά ξαφνικές ασκήσεις διασφαλίζουν πως, είναι, πως έχουν σε ετοιμότητα τις ένοπλες δυνάμεις τους. Ποια είναι η ιστορία αυτού. Δεν είμαι ειδήμων περιστρατιωτικών ζητημάτων. Δεν είμαι απλά δικηγόρος, αλλά από ό,τι θυμάμαι, από ό,τι γνωρίζετε το σύστημα, στην εποχή της Σοβιετικής Ένωσης χρησιμοποιούσαν πολύ έντονα τις ξαφνικές ασκήσεις. Την υψηλή ετοιμότητα των ένοπλων δυνάμεων αποτελούσε μέρος της στρατιωτικής εκπαίδευσης Πρόκειται λοιπόν για μια αναγέννηση του συστήματος αυτού με πολύ συστημικό τρόπο. Η άσκηση αυτή η Κάφκασος 2016 μας το έδειξε. Ήταν μια πολύ μεγάλη στρατηγική άσκηση που έλαβε χώρα το Σεπτέμβριο. Αλλά πιο πριν είχαν, μερικούς μήνες πριν είχαν ξαφνικές ασκήσεις. Τι κάνουν λοιπόν. Διασφαλίζουν πως οι στρατηγικές υποδομές που αλλάζουν επίσης πολύ γρήγορα Έχουμε και τον σχηματισμό των διάφορων πλατφορμών εντός των στρατιωτικών ομάδων. Κατάλαβαν λοιπόν πως πρέπει να είναι έτοιμοι όποτε χρειαστεί. Εάν σε δύο εβδομάδες από τώρα το, το ρωσικό καθεστώς, το οποίο από ό,τι ξέρετε δεν έχει μεγάλη κλίση προς τη δημοκρατία, μπορεί να αποφασίσει και να κάνει ό,τι θέλει. Καθώς όλα εξαρτώνται από έναν άνθρωπο, Οπότε λοιπόν τα στρατεύματά του είναι έτοιμα να κάνουν ό,τι θέλει. Δεν πρόκειται για μία απλόφα. Τα στρατεύματα όντω μπορούν να εφαρμόσουν αυτό που θέλει ο ένα άνθρωπο αυτό. Θέλουν λοιπόν να δημιουργηθεί αυτή η εικόνα μια διστακτική δύση, διστακτική να αναλάβει δράση, ακόμα και αν πρόκειται για σήματα ζωτικής σημασίας για τη δική της ασφάλεια και δυστυχώς ακόμα δεν είμαστε μέρος αυτής της ομάδας, αλλά τουλάχιστον οι χώρες που είναι μέλη του ΝΑΤΟ είναι επίσης στόχος της, της Ρωσίας. Θέλουν δηλαδή να μην αισθάνεται κανείς ασφαλής. Θέλουν να δημιουργήσουν έναν χώρο που δεν θα είναι πολυμερής. δεν είναι αυτό που εννοεί η Ρωσία όταν μιλάει για πολυπολικότητα. Είναι πολυπολικότητα του τύπου πως έχουμε πολλούς πόλους με δικά τους πεδία συμφέροντων χωρίς να επεμβαίνει κανείς και όπου ο καθένας κάνει τη δουλειά του όπως νομίζει. Και αν αυτό είναι ο κόσμο στον οποίο θα πρέπει να αποδεχτούμε να μένουμε, τότε θα πρέπει να ρίξουμε μια ματιά στην, στην Ασία. Επειδή στην Ασία και στην Νότιο Ασία, στην Νότιο Συνική Θάλασσα, μπορούμε ήδη να δούμε πού θα οδηγήσει ένα τέτοιο μοντέλο. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι ένα θέμα ζωτική σημασία για την ευρωπαϊκή ασφάλεια και την παγκόσμια ασφάλεια. Αυτή η έλλειψη τάξης, εάν δεν διατηρηθεί η διεθνή τάξη με κάποιο σεβασμό, τουλάχιστον κάποιο προ το διεθνές δίκαιο, με πονάει που το λέω, είμαι δικηγόρος με δίκευση στο διεθνές δίκαιο. Είναι δύσκολο πιστεύουμε, αλλά αυτό είναι το θεμέλιο μέσω του οποίου διατηρούμε την ειρήνη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και πιστεύω πως αξίζει να πολεμήσουμε γι' αυτό. Για μας είναι ζωτική σημασία τόσο για την Ουκρανία όσο και για τη Γεωργία. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε για το πάθος που δείχνετε στην παρουσίασή σας. Θέλω, Πρόεδρε και Πρέσβη, να σας ευχαριστήσω για τις συνελεχή παρουσία σας. Επειδή κανείς δεν ζητά το λόγο, θα ήθελα να ολοκληρώσουμε αυτό το σημείο και κλείνω με αυτή την πρόταση. Είστε εδώ διότι είμαστε πεπισμένοι ότι η επιβίωσή σας είναι προϋπόθεση για τη δική μας. Σημεριζόμαστε τις ανησυχίες σας για την ασφάλεια και γι' αυτό είσαστε εσείς εδώ και αντίστοιχα είμαστε παρόντες και εμείς στις χώρες σας και θα εξακολουθήσουμε σε αυτό το δρόμο. Θα αποχαιρετήσουμε τα μέλη του πάνελ θα κάνουμε μια τελευταία παρατήρηση. Okay. Ωραία, διάφορα. Πολύ πλούσια η, συνεδρίασή μας. Ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας. Η... Στις 12 ε, και 13 Οκτωβρίου θα γίνει η επόμενη συνεδρία. μας. Ευχαριστώ και πάλι για σήμερα. Αντίο.